Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε θερμά στην συνέχιση, στη συνεδρίαση αυτή για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Συνήθαν συναντήθηκαν ήδη από τις 9 στις 10 οι συντονιστές της Επιτροπής μας και για τις διάφορες αποφάσεις όπως ήθιστε γνωστοποιούνται αμέσως στη συνέχεια. Δύο σημεία έχουμε ακόμα από εχθές που ιστερότερα κατά τη διάρκεια του πρωινού θα τα εξετάσουμε εφόσον καταφέρουμε να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Στο σημείο 20 θα είμαστε στην προφορική ερώτηση δηλαδή της συναδέφου Αντωνέσκου Ελένα Τζοάννα Αντωνέσκου για τις ανισότητες όσον αφορά την επισητιστική ασφάλεια, την κάλυψη των επισητιστικών αναγκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστή η ερώτηση, το ζήτημα αυτό. Έχουμε τον κύριο Ζεγόμ Λεπέντρα από την ε, Γενική Διεύθυνση Αρμόδια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι δυνατόν να, του δώσουμε βέβαια τον λόγο, αλλά όταν θα έχουμε και την τεχνική που θα είναι έτοιμη θα έχουμε και μια ταινία τεσσάρων λεπτών που θα προβληθεί για αυτό το θέμα. Ο κύριος Λεπένθρα λοιπόν έχει τον λόγο. Θέλετε να μας ε, δώσετε τις πληροφορίες, να μας ενημερώσετε για αυτό το θέμα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τον Απρίλιο του 2011 έγινε μια έρευνα από Ένωση Καταναλωτών για μια σειρά τροφίμων, προϊόντων τροφίμων σε οκτώ κράτη-μέλη, όπου φάνηκε ότι στη σύνθεση των διαφόρων προϊόντων υπήρχαν αλλοιώσει, ανάλογα με τον τόπο εμπορία τους. Μάλιστα το ίδιο διαπιστώθηκε για τις συσκευασίες, ανάλογα με την ε, σύνθεσή του συσκευασιών. Περισσότερο από 200% μάλιστα. Η μελέτη των αποτελεσμάτων δεν μας δείχνει βεβαίως διαφορά στην ποιότητα μεταξύ των προϊόντων ανάλογα με το κράτος μέλος, αλλά περισσότερο στην ε, συσκευασία. Το, αυτό είσαι για τα σαχαρόδι ποτάλογου, χάρη με ισογλυκόζη. Εδώ, αυτό είναι ένα παράδειγμα προϊόντος που μπορεί να έχουμε υπόψη ανάλογα με τις συγκεντρώσει που παραγόνται σε λίγα εργοστάσια ανά τον κόσμο και μετά διατίθενται σε περισσότερα σημεία πώληση. Η τοπική αγορά για τα ποτά με ισογλυκόζη όπως ξέρετε ορίζεται από τους όγκους παραγωγής που διατίθενται στο εμπόριο. Η ζάχαρη χρησιμοποιείται στην Πολωνία και την Τσεχία από την άλλη. Δεν μιλάμε λοιπόν για διαφορές μεταξύ των ε, νέων και παλιών κρατών μελών. Η ισογλυκόζη χρησιμοποιείται πολύ σε διάφορα ποτά γιατί ακριβώς είναι πιο εύκολη η διάλυση του, στο ποτό. Στις Ηνωμένε Πολιτείες μάλιστα όπου υπάρχει η συνήθεια της κατανάλωσης ε, των ποτών αυτών, των soft drink, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο η ισογλυκόζη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις επιχειρήσεις λοιπόν να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις ε, ανάγκες των τοπικών καταναλωτών, τη διάθεση των πρώτων και την ε, συγκεκριμένη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να προστατεύσει την υγεία των καταναλωτών, σκοπό έχει να εγγυηθεί και την καλή λειτουργία τη ενιαία αγορά. Η βασική αρχή είναι ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην τοπική αγορά πρέπει να είναι υγιή. Οι καταναλωτέ να έχουν ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που καταναλώνουν. Είναι πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές για, τα, για τις ετικέτες των προϊόντων. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο σύντομα θα εγκρίνει το νομοθετικό πακέτο για να ενισχυθούν οι σχετικοί κανόνε. Επίση, θα πρέπει οι επιχειρήσει να προσαρμόζουν τα προϊόντα του στι διάφορε αγορέ. Η Νουτέλα, λόγω χάρη, μεταξύ Γαλλία και Γερμανία. Θα σα δείξω και το βίντεο, αν καταφέρουμε να το πετύχουμε το τεχνικό διακανονισμό. Υπάρχει διαφορά μεταξύ παλιών και νέων κρατών μελών. Θα πρέπει ο καταναλωτή να μπορεί να αποφασίζει ποιο προϊόν θα αγοράσει. Υπάρχουν φορές μεταξύ των διαφόρων ε, λογοτύπων και εμπορικών σημάτων. Αν ένας καταναλωτής δεν θέλει να αγορασει κοκακόλα θα στραφεί σε ένα άλλο προϊόν. Πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν και η ενημέρωση προς τον καταναλωτή, Ιδιώς με τη στήριξη των εθνικών ενώσεων καταναλωτών. Και ο Επιτροπός μας έχει δεσμευτεί να παρακολουθήσει το θέμα στενά. Voilà. Μάλιστα, πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Λεπέντρ. Θα δούμε τώρα το βιντεάκι, την ταινία. δεν γίνεται γιατί η τεχνική δεν είναι έτοιμη να την προβάλλουν. Εντάξει. Good, Ωραία, περνάμε στη συζήτηση. Αν σας κατάλαβα σωστά, μεριμνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υγεία, την υγιεινή αυτών των προϊόντων και τις σωστές πληροφορίες για την ενημέρωση των καταναλωτών, αλλά όχι για διακυμάνσεις και διαφορές των παραγωγών όσον αφορά την γεύση και τη σύσταση ενός προϊόντος. Συζητάμε τώρα αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Η Ελένα Αντωνέσκου παρακαλώ. Η ερώτησή σας ήταν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ήθελα όμως και εγώ με τη σειρά μου να παρατηρήσω κάτι. Δεν μιλάμε εδώ για προϊόντα τα οποία προσαρμόζονται στις διαθέσεις ή τις προτιμήσεις των καταναλωτών των διαφορετικών κρατών μελών. Όχι. Εδώ και αυτό ήταν το θέμα της ερώτησής μου, κάναμε λόγο για τη διαφορά στην ποιότητα μεταξύ προϊόντων που πολλούνται στα παλιά και στα νέα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή μας, ακριβώς γιατί ακόμα και αν δεν έχει υπάρξει μελέτη αυτή καθεαυτή, εμείς οι καταναλωτές βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ποιότητα, διαφορά στην ποιότητα των προϊόντων. Μέλη της οικογένειάς μου έχουν αγοράσει εδώ προϊόντα στις Βρυξέλλες, διότι θεωρούν ότι είναι ποιοτικό ανώτερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δύο κατηγορίες καταναλωτών, αλλά εάν αυτό αληθεύει είναι πολύ σοβαρό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δοκιμές που έγιναν από ενώσεις καταναλωτών στη Σλοβακία, η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να παραμείνει μόνο σε αυτά τα πειράματα και τις δοκιμές, να γίνουν και άλλες έρευνες. Εάν το πρόβλημα έχει ήδη διαπιστωθεί, αν άλλοι συνάδελφοι το έχουν παρατηρήσει και στο παρελθόν, νομίζω ο Υπουργό ε, Γεωργία τη Βουλγαρία το ανέφερε κάποια στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κινηθεί, να διεξαγάγει τι δικέ τη μελέτε, τι δικέ τη έρευνε για να δει αν υπάρχει διαφορά ποιότητα μεταξύ των προϊόντων που είναι αντικείμενο εμπορία στα διαφορετικά κράτη-μέλη τη Ένωση. Εάν αυτό ισχύει, είναι απαράδεκτη μια τέτοια κατάσταση. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Παύλ Πότς, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μείνω ήρεμο στο θέμα αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο καθώς πρέπει να μια από αυτές τις χώρες που θίγεται από το πρόβλημα και θα ήθελα να πω στην Επιτροπή ότι είναι η συμπεριφορά της απαράδεκτη. Μπορεί να φαίνεται σαν ίσονο σημασία πρόβλημα, αλλά δεν είναι. Και να σας εξηγήσω. Πρέπει να σας πω ότι κάθε μέρα ο κόσμος ε, θέτει τις ερωτήσεις, ενδιαφέρεται και ρωτάει όχι μόνο για τρόφιμα, αλλά ρωτάει ακόμη και πώς είναι δυνατόν να διατίθενται αυτά τα προϊόντα στην αγορά. Και μου λένε τι σημαίνει, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν μπορεί να μας προστατεύσει κατά αυτών των κακής ποιότητας προϊόντων. Πώ είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε την κρίση, μου λένε, πώ είναι δυνατόν να ανορθώσουμε την οικονομία μα, εάν μα ε, έχουν ξεχωρίσει έτσι και μα ε, υποβιβάζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα τρόφιμα, έχει μετατραπεί σε ένα πολιτικό πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο εθνικέ κυβερνήσει, αλλά μεγάλε και ε, πολυεθνικέ επιχειρήσει. Δεν πρέπει λοιπόν να δείχνουμε υποχωρητικότητα, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Δεν αρκεί να μιλάμε πια, έχει τελειώσει η εποχή που μιλάγαμε, τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τσάμπα βάζει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω την προσοχή των συναδέλφων να την στρέψω στο ότι εμείς πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, πολύ προσεκτικοί. Και εγώ προέρχομαι από ένα νέο κράτος μέλος, διότι ακόμα και οι δοκιμές των σλοβακικών πειραματικών δικαστη... Ε, εργαστηρίων δεν είναι με εμφανή αποτελέσματα. Για παράδειγμα στην Coca-Cola δεν μπορούσαν να βρουν τη διαφορά μεταξύ παλαιών και νεότερων κρατών μελών. Πρόκειται λοιπόν το για το θέμα της ισογλυκόζης και της χρήσης της στη Σλοβακία, Ρουμανία, Βουλγαρία και σε άλλα περαιτέρω κράτη-μέλη η Coca-Cola γλυκαίνεται, χρησιμοποιεί τον, την γλυκαντική ουσία ισογλυκόζη, ενώ αλλού την σακχαρόζη. Δεν πρόκειται για το ότι ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει πάντα μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Όμως θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους αυτό να μην το θεωρήσουν λαϊκισμό, πολιτικό λαϊκισμό και έτσι ότι γίνεται κάποια κατά, ε, κατάχρηση. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση η υγιεινή των τροφίμων, το θέμα των υγιεινών τροφίμων. Για το θέμα της δικής μας δραστηριότητας εδώ πρόκειται και για αρμοδιότητα και της Επιτροπής ΙΝΚΟ. Θα έπρεπε από την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή να συνεργαστούμε και να δούμε και ποια είναι η αναλογία σε σχέση με τις τιμές, διότι όταν υπάρχει διαφορετική ποιότητα σε ένα προϊόν θα πρέπει να αντανακλάται η διαφορετική σύνθεση και ποιότητα και στις τιμές. Και ένα άλλο περαιτέρω στοιχείο που αναφέρθηκε είναι ότι υπάρχει αρνητική διακριτική μεταχείριση λόγω όλων αυτών των στοιχείων. Λοιπόν και στην Ουγγαρία υπήρξαν δοκιμές που έγιναν και αυτές οι εξετάσεις ε, που έγιναν μόνο μερικά, μόνο εν μέρη επιβεβαίωσαν τις, ε, τα πειράματα στη Σλοβακία, αλλά υπήρχαν και άλλα προϊόντα, όπως ε, για παράδειγμα οι πάνες των μωρών, όπου υπήρχαν τεράστιες διαφορές όσον αφορά την απορροφητικότητα αυτών των πανών. Μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις πάνες που πουλούσαν στην Αυστρία και άλλες που ήταν διαθέσιμες και επολούντος στην Ουγγαρία και η Επιτροπή μας σε σχέση με τα θέματα της υγιεινής τροφίμων δεν έχει την κύρια αρμοδιότητα. Όμως η υγεία των καταναλωτών που πρέπει να προστατευτεί είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Και οι δύο μας επιτροπές, Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καταναλωτών πρέπει να συνεργαστούν διότι και οι δύο πτυχές πρέπει να συνεξεταστούν. Και θα ήθελα να πω ότι την συνάδελφο από ε, τους άλλους συναδέλφους τους κατανοώ σε αυτά τα οποία είπαν. Θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω εξετάσεις αλλά επιστημονικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Άντερ παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, δεν είναι σύμπτωση ότι και οι τρεις παρεμβάσεις προήλθαν από χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης. Επίσης δεν είναι σύμπτωση δεν είναι τυχαίο ότι εμείς όλοι αμέσως αντιδράσαμε σε σχέση με αυτές τις ειδήσει, διότι αφορά η ερώτηση αυτή τη συναδέλφου από τη Ρουμανία ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο από την Ουγγαρία. Πρόκειται για την ασφάλεια των τροφίμων, για την προστασία των καταναλωτών και για θέματα ανταγωνισμού. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σύνθετο περίπλοκο ζήτημα. Η δήλωση που ακούσαμε δεν μπορεί να γίνει δεκτή η τοποθέτηση που ε, μας εξέθεσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Η ε, επιχειρήσεις για την σύνθεση των προϊόντων τους ότι θα πρέπει λέει να προσαρμόζουν τα προϊόντα αυτά στη γευστικά και όσον αφορά και την τιμή τους ε, η ποιότητα δεν είναι ε, το κυριότερο θέμα εδώ όσον αφορά αρνητικές πτυχές της αλλά η σύνθεση είναι διαφορετική ούτως ή άλλως και γι' αυτό σε σχέση με τα θέματα της κυρίας Αντωνέσκου είναι, σαφή αυτές, είναι σαφείς αυτές οι πτυχές. Είχαμε ένα προϊόν και εδώ κάνω λόγο εγώ μόνο για τρόφιμα είναι η, το, η σοκολάτα Μίλκα αλλά δεν υπήρχε ούτε ένα άλλο προϊόν όπου στην ε, Ευρώπη και στην κεντροανατολική Ευρώπη να υπάρχει ε, κάποια διαφορά. Εδώ στην ε, στις Βρυξέλλες όταν πηγαίνω σε ένα κατάστημα την ίδια σοκολάτα μίλκα μπορώ να αγοράσω όπως στην Ουγγαρία. Όμως τα άλλα προϊόντα δεν συμβαίνει αυτό. Στην Πράγα και στην Βουδαπέστη αγοράζει κανείς προϊόντα που έχουν τελείως διαφορετική ποιότητα και σύνθεση από ότι εκείνα που αγοράζει στο Παρίσι. Γι' αυτό αυτή η ερώτηση. Κάποιοι παραγωγοί, όχι όλοι, αλλά κάποιοι συγκεκριμένοι παραγωγοί παραδέχτηκαν, ομολόγησαν ότι φθηνότερες ε, ουσίες, συστατικές ουσίες χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή των προϊόντων τους ε, στην κεντροανατολική Ευρώπη. Και εδώ είναι η ουσία του πράγματος, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί ομολόγησαν ότι χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν φθηνότερα συστατικά για την παραγωγή των προϊόντων τους. Και όταν έχουμε και την διαμόρφωση των τιμών, για παράδειγμα στις αγορές ε, της κεντροανατολικής Ευρώπης, ξέχασαν εντός εισαγωγικών, ξέχασαν να ενημερώσουν τους καταναλωτές για το Οι διαφημίσεις ήταν ακριβώς οι ίδιες, πανομοιότυπες, τα προϊόντα ήταν τα ίδια υποτίθεται, αλλά η ποιότητά τους ήταν τελείως διαφορετική και πολύ, πολύ χαμηλότερη η ποιότητά τους, υποβαθμισμένη και έτσι εισέπραταν υπερβολικό κέρδος το οποίο ενθυλάκωναν πουλώντας αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν ήταν ε, η, ε, η ίδιας ποιότητας και σύνθεσης με εκείνα ε, που διέθεταν στην Δυτική Ευρώπη. Τώρα, αν υπάρχουν αμφιβολίες ή αν χρειάζονται περαιτέρω αποδείξεις, λέει κάποιος, οι σλοβακικές πειραματικές ενέργειες αν θέλουμε να συμπληρωθούν ή να επεκταθούν αυτά τα πειράματα, θα πρέπει άμεσα να αντιδράσουμε για να γίνει κάτι. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Πότς. Σε σχέση με όλα αυτά έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. χρόνος πιέζει ασφικτή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα έπρεπε αυτά τα πειράματα το δυνατόν πιο γοργά να τα διεξαγάγουν και οι πιο αυστηρές κυρώσεις και ποινές θα πρέπει να επιβληθούν σε περίπτωση παραβιάσεων. Παρακαλώ εσείς έχετε τον λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάιμες θα ήθελα να πω ότι προσέχω ότι εδώ πρόκειται για ένα παλαιό, πολύ παλαιό φαινόμενο ουσιαστικά για την κρίση του τι εστί ποιότητα. Η ποιότητα εξαρτάται μόνο από την τιμή ή εξαρτάται και από κάποιους άλλους συντελεστές, από κάποιες άλλες παραμέτρους. Όταν κάτι είναι φθηνότερο ποιοτικά είναι υποβαθμισμένο και χειρότερο, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα συνεξετάσουμε. Είμαι Γεωργός και στην χώρα μας για παράδειγμα ε, πρέπει να δούμε ότι στα λιβάδια μας, ε, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν ε, ε, κάποια, ε, κάποιες χορτολιβαδικές εκτάσεις όπου έχουμε καλύτερο χόρτο, όπως ε, μπορεί όμως και στο γειτονικό χωράφι να διαπιστώνεται ότι για τις αγελάδες ε, υπάρχουν και ε, αντικειμενικά κριτήρια γιατί είναι πιο γευστικό το χορτάρι σε, ε, κάποια, σε κάποιες εκτάσεις, σε κάποια χωράφια. Αυτό πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, γιατί όταν κατηγορούμε τις εταιρείε ότι θέλουν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην σύνθεση ενός προϊόντος δεν έχουμε ακριβώς τις ίδιες ποσότητες και την ίδια σύνθεση παράδειγμα για τις μαρμελάδες από φράουλα. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες μαρμελάδες, ε, οι ίδιες φράουλες που, χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται ε, οι φράουλες αλλά που από πλευράς ποιότητας ή από πλευράς ε, συστατικών που προστίθενται δεν είναι ακριβώς ε, στο τελικό προϊόν η ίδια η ποιότητα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη εδώ αν υπάρχει ενέργεια η οποία υποκρύπτει κάποια παραπλάνηση ή αν όλα αυτά οφείλονται στις μεθόδους παραγωγής και στη σύνθεση των προϊόντων για την χρήση για παράδειγμα κάποιων συστατικών ουσιών που θα ε, χρησιμοποιούσαν κάποιες εταιρείες. Όλα αυτά πρέπει ανοιχτά και ειλικρινά να τα συζητήσουμε με τις παραγωγούς εταιρείες και να μην προδικάζουμε το τι συμβαίνει. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα νομικές δυνατότητες διαθέτουμε για να ρυθμίσουμε τη σύνθεση και τα συστατικά, τις συνταγές που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείε. Εδώ έχουμε συγκεκριμένε περιπτώσεις, μιλάμε για μια συγκεκριμένη κατάσταση και ακούσαμε να προβάλλονται διαφορετικά επιχειρήματα. Ένα συνάδελφος μόλις είπε ότι διαφορετικά συστατικά χρησιμοποιούνται από χώρα σε χώρα. Λόγω χάρη στον χυμό πορτοκαλιού, πορτοκαλάδα. χρησιμοποιούνται πορτοκάλια από διαφορετική, διαφορετικής προέλευσης. Όμω, ε, αυτό πρέπει να έχουμε επίση υπόψη είναι ότι είναι διαφορετική αγοραστική δύναμη των καταναλωτών από μέρο σε μέρο. Άρα, ε, κάποια συστατικά αντικαθίστανται από άλλα φτηνότερα. Υπάρχει λοιπόν νομική δυνατότητα να διευθετήσουμε το θέμα των συνταγών που χρησιμοποιούνται από τι εταιρείε. Τελευταία παρέμβαση της κυρίας Άννα Ρόσμπαχ, παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω δανέζικα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι σκάνδαλο αυτή η κατάσταση. Προέρχομαι από μία από τις δυτικές ε, χώρες μέλη και βλέπω όλο και περισσότερο δυτικοευρωπαϊκές εταιρείες που μεταθέτουν την παραγωγή τους στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά και έχουμε την ελευθερία κυκλοφορίας των αγαθών και είναι κάτι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς, δεν μπορώ εγώ να το κατανοήσω γιατί οι δυτικοευρωπαϊκές βιομηχανίες οι οποίες μεταθέτουν την παραγωγή τους στην Ανατολική Ευρώπη για παράδειγμα όσον αφορά τις μαρμελάδες ε, φράουλας ε, ή ε, όσον αφορά και τα πορτοκάλια, γιατί χρησιμοποιούν διαφορετικές συνταγές. Μια και υπάρχει ελευθερία κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν πιο προσεκτικά σε βάθος αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες αγαθών, πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, ενώ παράγονται από τις ίδιες βιομηχανίες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε οπωσδήποτε με ιδιαίτερη προσοχή. Ίσως για παράδειγμα όταν αγοράζει κανείς κάποια προϊόντα αναβαθμισμένα ή υποβαθμισμένα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε τις ίδιες εταιρείε που παράγουν στην Ανατολική Ευρώπη και μεταφέρουν και πολλούν αυτά τα προϊόντα τους και στη Δυτική Ευρώπη. Πρέπει αυτό να το θεωρήσουμε απαράδεκτο και πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος με προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν ε, μεγάλες ευαισθησίες ε, που θίγονται και πολύ μεγάλες, ε, μεγάλο ενδιαφέρον και μέλημα να μην προσφέρουν διαφορετικής ποιότητας προϊόντα, όχι μόνο διαφορετικής, γευστικής, γε, διαφορετικής γεύσης προϊόντα, αλλά και διαφορετικής ποιότητας και καμιά φορά με υψηλότερο αντίτιμο, υψηλότερη τιμή η Επιτροπή μας θα πρέπει να ρωτήσει αν υπάρχει μία μείωση της ασφάλειας τροφίμων σε σχέση με αυτό το θέμα. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να κληθεί να συντάξει περισσότερες μελέτες και να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τη μία ή άλλη χώρα και για τη διαφορετική σύσταση των προϊόντων αυτών και να δούμε αν υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια, επιστημιστική ασφάλεια αυτών των τροφίμων. Κάτι άλλο ως θέμα είναι η παραπλάνηση των καταναλωτών. Αναφέρθηκε από πλευρά συναδέλφου ότι το ίδιο προϊόν με την ίδια ετικέτα, με την ίδια διαφήμιση έχει διαφορετικές συστατικές ουσίες στη σύνθεσή του. Τίθεται το ερώτημα, είναι παραπλάνηση των ε, καταναλωτών αυτών, παραβιάζονται κάποιες αρχές ε, του δικαίου ανταγωνισμού. Τώρα να συντάξω μια επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Επιτροπής ε, ΙΝΚΟ ως ε, Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών να υπάρξει ε, προσπάθεια συνεξέτασης αυτού του θέματος. Θα πρέπει να εξεταστεί και από αυτούς αυτό το θέμα. Τώρα τέθηκε ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν νομικές δυνατότητες να ελέγχουμε τα τις συστατικές ουσίες συνταγών παραγωγής τροφίμων Υπάρχει δυνατότητα να γίνεται αυτό. Θα συντάξει περαιτέρω μελέτε για αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε και το βιντεάκι των τεσσάρων λεπτών διάρκεια που ε, ήθελατε να μα προβάλλετε. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την ε, νομοθεσία, κοινοτική νομοθεσία για τα τρόφιμα, εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την υγεία του καταναλωτή, αλλά δεν μπορεί να περιγράψει το, τα συστατικά των τροφίμων. Δεν μπορούμε δηλαδή να διανοηθούμε ότι θα ε, υπαγορεύουμε τη χρήση του τάδε ή του δίνα γλυκαντικού. Τα πρόσθετα είναι μια άλλη ιστορία γιατί είναι ζήτημα υγείας, αλλά δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή ειναι ζητημα υγεια αλλα δεν μπορει η ευρωπαικη επιτροπη να επιβάλλει συνταγή για τα τρόφιμα που διατίθεται στην αγορά. Ένα άλλο ζήτημα είναι η δύναμη του που έχει ο καταναλωτή. Εάν ο καταναλωτή βρίσκει ότι ένα προϊόν δεν είναι ικανοποιητική ποιότητα, θα στραφεί προ άλλο προϊόν. Άρα δεν πρέπει να υποτιμούμε την ισχύ, τη δύναμη που έχει ο καταναλωτή. Τα κράτη-μέλη από την άλλη έχουν επίση ρόλο ελέγχου τη τήρησης τη κοινοτική νομοθεσία, δηλαδή ότι τα προϊόντα που διατίθεται στην αγορά είναι ευθυγραμμισμένα με την κοινοτική νομοθεσία. Και φυσικά θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ιδιαίτερη προσοχή θα παρακολουθεί στην εξέλιξη του θέματος αυτού και ιδιαίτερα στο τομέα της ε, βελτίωσης της ενημέρωσης του καταναλωτή. Αυτό είναι το βίντεο το οποίο ήθελα να σας δείξω, την ε, σχέση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, δύο παλαιών κρατών δηλαδή, όπου με το ίδιο προϊόν, την ίδια ετικέτα, το ίδιο ε, την ίδια συσκευασία έχει διαφορετική σύνθεση το προϊόν, μόνο και μόνο για να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις αγοράς. Στην ίδια ε, χώρα μέλος υπάρχουν διαφορές ακόμη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Γαλλίας. Από ό,τι ακούω είναι διαφορετικό το ποσοστό της ζάχαρης στα σοκολατούχα προϊόντα, γιατί έχει προσαρμοστεί η αγορά στις προτιμήσεις του καταναλωτή. Να σας δείξω τώρα, αν μου επιτρέπετε, αυτό το βίντεο που δείχνει τις αποκλήσεις.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 Και όταν κάνει ο Γερμανός φίλος μας το ίδιο πράγμα με τη γερμανική νουτέλα σε μια γερμανική φέτα ψωμί, για κοιτάξτε πώς μασούν και γεύονται την φέτα με την νουτέλα, πραγματικά γεμίζει σάλια το στόμα από την όρεξη να φάει και, κανείς το ίδιο. Και τώρα αλλάζουν τα κουτιά, το γερμανικό κουτί πάει στην Γαλλία και αντίστροφα. Τώρα παίρνει καθένας μια νέα φέτα ψωμί και την αλήθει πάλι με νουτέλα. Και τι βλέπει, στην γερμανική πλευρά όλα είναι τέλεια. Ο φίλος <clears throat> χρησιμοποιεί το, τη γαλλική νουτέλα στη φέτα του. Για να δούμε τι κάνει τώρα ο Γάλλος με τη γερμανική νουτέλα. Όπως βλέπετε εδώ προφανώς υπάρχει μια ασυμβατότητα μεταξύ γαλλικού ψωμιού και γερμανικής νουτέλα ασυμβατότητα, μια και είναι πιο παχύρευστη η νουτέλα αυτή. Ο Γάλλος φίλος μπορεί να προσπαθήσει όσο και αν θέλει, αλλά το ψωμί του αυτό διαλύεται και καταστρέφεται η φέτα του αυτή. Η νουτέλα δεν ταιριάζει σε αυτό. Καταστροφή όλεθρος. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε οπωσδήποτε ότι δεν έχουν την ίδια ε, σύσταση η γαλλική νουτέλα και η γερμανική νουτέλα. Πρόεδρος, πολύ ωραίο σλάπστικ αυτή η ταινία που είδαμε. Και επεξηγεί ίσως και γιατί η γεύση από χώρα σε χώρα και σε μεγάλες χώρες και όλα και του Βορρά ή του Νότου έχουν διαφορές. Αλλά αυτό δεν ήταν ακριβώς το θέμα μας. Το θέμα μας είναι η ποιότητα. Και έτσι μέσω της ποιότητας η ασφάλεια των τροφίμων. Και έτσι για την Επιτροπή ΙΝΚΟ ίσως και η παραπλάνηση των καταναλωτών και τι συμβαίνει σχετικά. Λοιπόν, τα είδαμε, τα συζητήσαμε. Εγώ θα συντάξω και θα αποστείλω μια επιστολή στο Μάκομ Harbor ώστε η δική του Επιτροπή ΙΝΚΟ να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες και τεκμήρια. Ίσως να ζητήσετε να συνταχθεί μια μελέτη, όχι μόνο όσον αφορά τις γευστικέ διαφορές αλλά όσον αφορά και τις πραγματικές αυθεντικές ποιοτικέ διαφορές που αγγίζουν και στα όρια της ασφάλειας τροφίμων τουλάχιστον μπορεί κανείς να δει ότι με χαμηλότερη ποιότητα ζητούν και απαιτούν υψηλότερο αντίτιμο, υψηλότερη τιμή. Θα πρέπει να δούμε ότι βλάπτονται οι καταναλωτές με αυτό, τον τρόπο, με αυτό το κόλπο. Δεν πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε με κάτι τέτοιο, να υπάρχουν επιπλέον κέρδη μέσω μιας τέτοιας διεργασίας, εσχροκέρδειας δηλαδή, δεν θα το δεχόμαστε αυτό. Να ολοκληρώσουμε με αυτό το θέμα γιατί πιέζει και η ημερήσια διάταξη. Ευχαριστούμε για την ερώτηση που θέσατε γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν διαμαρτυρίες, ανασφάλεια, αβεβαιότητα και δεν μπορεί να δεχθεί το Ευρωκοινοβούλιο μια τέτοια κατάσταση βέβαια. Ναι. Αν και ανησυχώ ότι τελικά ήταν περισσότερο διαφημιστικό το φιλμάκι που είδαμε παρά διαφωτιστικό. Εάν λοιπόν καλά κατάλαβα, βάσει της ε, παρουσίαση τη Επιτροπή, μα λέει η Επιτροπή ότι έχουν το δικαίωμα οι εταιρείε να προσαρμόσουν τη σύνθεση των προϊόντων τους, ανάλογα με τι τοπικέ προτιμήσει ή ανάγκε, ε, αρκεί να σέβονται την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τέλο πάντων, δεν υπάρχει λοιπόν ευρωπαϊκό νόμο για να τιμωρηθεί η διακριτική μεταχείριση των καταναλωτών. Να πω λοιπόν και εγώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσω έπρεπε να το σκεφτείτε αυτό. Να σα απασχολήσει το θέμα εφ' εξής. Περιμένουμε να δούμε και μια πρόταση από εσά βάσει πρόσθετων μελετών και στοιχείων, διότι οι ενώσει καταναλωτών που εκπροσωπούν τα διαφορετικά κράτη-μέλη μας το έχουν επισημάνει το θέμα. Περιμένω λοιπόν να προταθούν και λύσεις. Ευχαριστώ. Καλώ. Καλώς. Η Επιτροπή άκουσε τι έχουν να πούν τα μέλη της Επιτροπής, τι σκέφτονται, τι ζητούν. Θα επανέλθουμε φυσικά στο θέμα. Ίσως να έχετε και νέα στοιχεία εντωμεταξύ στους επόμενους μήνες και να μπορείτε να μας ενημερώσετε. Βλέπετε ότι υπάρχει πράγματι ανησυχία ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που υποβαθμίζεται μερικές φορές ανάλογα με το κράτος μέλος. Και περνώ στο επόμενο θέμα της ημερησής διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης πολύ ενδιαφέρον και συναρπαστικό. Εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων. Καταγωγή ή προέλευση Ιαπωνία μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό τη Φουκουσίμα. Όλοι παρακολουθήσαμε την τραγωδία αυτή και την εξέλιξη στον τομέα των, της εξέλιξης μας στον τομέα των, ρυθμίσεων, των εισαγωγών από την Ιαπωνία. Εγώ είχα σπεύσει να, προσ... συζητήσω με τον πρέσβη της ε, Ιαπωνίας, ο οποίος είχε διαμαρτυρηθεί την εποχή εκείνη για αρνητική ε, διάκριση εις βάρος των προϊόντων από την Ιαπωνία. Ας δούμε ποια είναι η κατάσταση. Έχουμε τον κύριο Βλατίσλαφ Μίκο, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, προστασίας υγεία του καταναλωτή και το Φραν Στρέτερ που θα μα πούνε τι ισχύει, τι συμβαίνει. Ο κύριο Μίκο έχει το λόγο πρώτο. Καλημέρα σα. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκινώ λέγοντας ότι είναι όντως ένα πολύ λεπτό όσο και ευαίσθητο θέμα. Το παρακολουθούμε στενά, καθημερινά. Ο λόγος για τον οποίο το συζητούμε είναι μεταξύ άλλων το γεγονός ότι ε, ο κύριος Λάινεν μας επέστειλε μια επιστολή ρωτώντας μας ε, να δώσουμε εξηγήσεις γιατί καθυστερήσαμε ως προς την ενημέρωση περί παράτασης των μέτρων. Ομολόγω ότι όντως δεν είχαμε αρκετό χρόνο να επαληθεύσουμε, να ελέγξουμε τα προτινόμενα, αλλά προσπαθούμε πάντοτε να ακολουθούμε τους κανόνες και να δίνουμε πληροφορίες ακριβώς την ίδια εποχή που τις προσφέρουμε και στα κράτη-μέλη. Ο λόγος της καθυστέρησης είναι ότι έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση που αλλάζει, που εξελίσσεται καθημερινά. Περιμέναμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα αναλύσεων ε, από την Ιαπωνία, τα οποία τώρα ελέγχουμε, τα παρατηρούμε και θα περιμένουμε την απόφαση επί τη βάση των πιο πρόσφατων πληροφοριών και εξελίξεων ε, από την Ιαπωνία. Εδώ λοιπόν εγώ βρίσκομαι για να σας δώσω πρόσθετες εξηγήσεις και να επισημάνω ότι θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθούμε πάντοτε στο μέλλον να σας ενημερώνουμε το ταχύτερο δυνατό. Αλλά αντιλαμβάνεστε πιστεύω ότι όταν ε, έχουμε να κάνουμε με την άρση ή την παράταση αυτών των σημαντικών μέτρων, το μόνο που μπορούμε να πράξουμε είναι να ακολουθήσουμε το δυνατόν πιο πρόσφατες και επίκαιρες πληροφορίες. Και άρα εξαρτώμαστε από τις εκκρίμεις ακόμη στην Ιαπωνία αναλύσεις. Θα σας ενημερώσω επίσης για κάτι που μάλλον γνωρίζετε, ότι η μόνιμη επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου ομόφωνα ε, ενέκρινε την παράταση των υφισταμένων μέτρων μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Ήδη έχουν τεθεί δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου σε ε, ισχύ αυτές οι αποφάσεις, οι αποφάσεις περί Έτσι είμαστε καλυμμένοι γιατί τα προηγούμενα μέτρα ισχύαν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Είμαι ικανοποιημένο γι' αυτό λοιπόν, διότι όπως βλέπετε είχαμε πίεση χρόνου πάνω απ' όλα να μην καθυστερήσουμε έτσι ώστε να, ε, και να μην υπάρξει κενό στην εφαρμογή των μέτρων. Επίσης βέβαια θέλουμε να δώσουμε στο δυνατόν πιο ικανοποιητική απάντηση στις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις σας. Ξέρετε ότι η παράταση υιοθέτηθηκε με ορίζοντα μέχρι τα τέλη του έτους αλλά με μηνιαία αναθεώρηση άρα έχουμε πολλές δυνατότητες να ανταποκριθούμε στις οποίες εξελίξεις και επίσης θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να σας δώσω κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τα μέτρα που έχουμε τώρα ενισχύει. Τι προβλέπετε λοιπόν. Τα μέτρα που έχουμε ενισχύει προβλέπουν ότι ζωοτροφές και τρόφιμα που προέρχονται από 12 ε, επαρχίες ή νομούς καλύτερα της Ιαπωνίας ελέγχονται πριν από την εξαγωγή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, παρουσία ιωδινίου 1.31, συνθεσίου 1.34 και συνθεσίου 1.37 και με πιστοποίηση ότι δεν έχουν ε, επίπεδα τέτοιων ε, μορίων, ραδιναργών μορίων και επίσης για 10 ακόμη νομούς έξω από τους 12 γίνονται ε, και άλλοι έλεγχοι. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα μέτρα τα ευρωπαϊκά που επιβάλλονται αυτή τη στιγμή για τις αγωγές ζωοτροφών και τροφίμων από την Ιαμπονία και ότι δεν έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλες ποσότητες, στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και είναι κατά την έποψή μας αναλογικά ως προς την ε, ποσότητα και τον κίνδυνο ε, και έτσι είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων από την Ιαπωνία. Θα ήθελα επίσης να δώσω επιπλέον πληροφορίες για τις εξελίξεις τις σχετικές με τις επιμέρους επαρχίες της Ιαπωνίας, καθώς πρόκειται για μια μάλλον ιδιάζουσα κατάσταση. Έχουμε τη Σουζιόκα επιπλέον προσθέσει ως επαρχία μετά το ε, ατύχημα που ξέρετε το, έγινε τον Ιούλιο διότι η έλεγχοι, οι επαληθεύσεις που έγιναν από την κυβέρνηση Ιαπωνίας σημειώνουν υψηλή συγκέντρωση αραδιενεργών σε προϊόντα πράσινου τσαγιού, που μπορεί με να είναι μικρή ποσότητα, αλλά από την άλλη έχει μεγάλη εισαγωγή, στην, μεγάλες ποσότητες εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουμε την ε, Άνια Μάγκατα και τις δύο αυτές επαρχίες που ελέγχθηκαν τα προϊόντα τους ε, και απεδείχθησαν καθαρά και έτσι βγήκαν από τον κατάλογο των ε, περιορισμών τον Ιούλιο. Ιδιαίτερη προστασία έχουμε επίσης δείξει για τη συγκέντρωση ραδιενεργού κεσίου σε ε, προϊόντα βοήου κρέατος και ενώ δεν υπάρχουν εξαγωγές βοήου κρέατος, εμείς παρακολουθούμε και πάλι την κατάσταση, έχουμε επακριβείς πληροφορίες για την Ιαπωνία και μας έχουν δοθεί εξηγήσει ότι η επιμόλυνση αυτή έχει να κάνει με τη χρήση κυρίως τροφών επιμολυσμένων ε, με ραδιενεργά, ε, και κυρίως ε, βλαστών ε, του φυτού της όριζας. Άρα όλα αυτά δεν αφορούν εμάς γιατί δεν επιτρέπεται η εξαγωγή βόηου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους δημόσιας υγείας και για λόγους υγείας των ζώων και όχι για λόγους ραδιενεργού επιμόλυσης. Πάντως επειδή απεδείχθη ότι δεν σχετίζεται με τις τοπικές επιμολύνσεις, οι ε, διαπιστώσεις αυτές ε, υπάρξης και σίου στο Βόλιο Κρέας δεν οδήγησαν σε παράταση, των, σε επέκταση μάλλον των μέτρων. Κατά τα άλλα συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν τακτικά την παρουσία αυτών των τριών ραδιενεργών ε, μορίων που ανέφερα νωρίτερα και στον τομέα των ψαριών από τις ζώνες FAO 5167 77 τα αλλιευόμενα ψάρια και προϊόντα ε, χθιοτροφίου πρέπει να επαληθεύονται. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι παρακολουθούμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων των εισαγωγών, τα οποία μέχρι τώρα ε, επιδεικνύουν μια πολύ θετική εικόνα ως προς τα επίπεδα των επιμολύνσεων ε, ζωοτροφών και τροφίμων που εισάγονται από την Ιαπωνία. Εκτός από δύο μερίδες πράσινου τσαγιού δεν εντοπίστηκαν ραδιενεργά, απόβλητα, ραδιενεργά ίχνη μάλλον και όπου υπήρχαν ε, ίχνη ραδιενέργεια ήταν ακόμη χαμηλά σε σχέση με το όριο. Πάντως εμείς συνεχίζουμε τις, ε, τους ελέγχους μας και τους δημοσιεύουμε στην ε, ιστοσελίδα μας για να είναι προσβάσιμοι στο κοινό. Παρακολουθούμε εκ του σύνεκης εκ Επιτροπή Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κατάσταση και αν χρειαστεί θα λάβουμε αμέσως τα απαραίτητα, τα πετούμενα μέτρα. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω, να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν και κάποιες προσπάθειες με μοντέλα στην Ιαπωνία να διαγνωστούν πιθανά ή πιθανολογούμενα προβλήματα σε άλλες περιοχές και αυτά τα παρακολουθούμε επίσης. Άρα εάν κάποιο μέχρι τώρα δεν είναι γνωστό φανεί ότι ενδέχεται να υπάρχει, θα αντιδράσουμε αμέσως. Και πριν κλείσω θα ήθελα να επισημάνω στατιστικά στοιχεία για την ενημέρωσή σας, στατιστικά στοιχεία που είχαμε προβλέψει για μια προηγούμενη συνεδρίαση που ακυρώθηκε όμως λόγω εκείνου του προβλήματος με το ηλεκτρικό ρεύμα. 1222, 1222 έλεγχοι που έχουν καταγραφεί από τα κράτη-μέλη, εκ των οποίων 909 για ζωοτροφές ε, και τρόφιμα από την Ιαπωνία και 313 από την υπόλοιπη ζώνη του ειρηνικού, δηλαδή προϊόντα ηχθείων, αλλά όχι από την Ιαπωνία. Πέραν αυτών των δύο περιπτώσεων στο πράσινο τσάι που σας ανέφερα δεν υπήρχαν ε, ποσότητες ανώτερες από το επιτρεπόμενο όριο ραδιενεργών ουσιών. Σε κάποιες μία που υπήρχε κάποια ε, ε, ίχνη ραδιενεργών ήταν πάντα κάτω από το όριο. Έχουμε μια-δύο περιπτώσει ε, και ΣΥΟ 1.34-1.37 σε πολύ μικρέ ποσότητε. Πάλι δεν υπήρχε θέμα δηλαδή μη τήρηση ε, των ορίων. Μία ή δύο περιπτώσει κατά πολύ λίγο είχαμε υπέρβαση με ραδιενεργή, ε, παρουσία ραδιενεργού ουσίας, ραδιενεργού ουσίας, αυτή ήταν πριν από την επιβολή των μέτρων. Και όσο και τη στιγμή που έχουν τεθεί τα μέτρα και εφαρμόζονται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα παράβασης και υπέρβασης. Και θα ήθελα κλείνοντα να αναφερθώ στα φυστάμενα μέτρα που παρατείνονται, όπως σας είπα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η στο επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων, με βάση βέβαια τα επιστημονικά στοιχεία και με την ε, αρχή τη αναλογικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισήγηση και για την υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μελλοντικά έγκαιρα, ενωρίς να μας πληροφορεί, να μας ενημερώνει σχετικά. Έχουμε και εκπροσώπους της ε, ε, Ιαπωνικής ε, Πρεσβείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε τον επικεφαλής και τους συναδέλφους του. Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση και στην Ευρώπη και παγκόσμια για αυτόν τον τεράστιο σεισμό που έπληξε και τα θύματα που υπήρξαν στην Ιαπωνία και το πυρηνικό ατύχημα στο σταθμό της Φουκουσίμα έχει πολύ μεγάλη υψηλή παράδοση όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων και τα σχετικά θέματα η Ιαπωνία. Παρόλα αυτά θα κατανοήσετε ότι οι πολίτες μας πρέπει να μεριμνούν και να προστατεύονται σε σχέση με τρόφιμα τα οποία αναφέρεται ότι είναι μολυσμένα. Ακούσαμε την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 220 δειγματοληπτικές τέτοιες έρευνες σε κάποιες τέτοιες ε, εξετάσεις και για τα τέλη Δεκεμβρίου 2011 που θα λήξει αυτή η περίοδος αν δεν υπάρξει άλλη απόφαση κτλ. Έχουμε συναδέλφους που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Ο Κρήτον Ασένης πρώτος, παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εφόσον βρισκόνται εδώ εκπρόσωποι της Ιαπωνικής κυβέρνησης, ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου για το γεγονός ότι θα συνεχίσει τη φαλαινοθυρία. Η Ιαπωνία. Και εν ώψη του μέλλοντος και μετά τα καταστροφικά γεγονότα στην ε, Ιαπωνία. Βρισκόμαστε στο πλευρό της Ιαπωνίας, αλλά δεν θέλουμε να προβλέψουμε και ανάλογα μέτρα. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ιαπωνία και όχι να την τιμωρήσουμε. Έχω μια σειρά ερωτημάτων, λοιπόν, οποία, τα οποία απαντήθηκαν από την Επιτροπή. Μάλλον θα πρέπει να συνεχίσουμε να ερευνούμε τον κίνδυνο που μπορεί να προέρχεται από τα προϊόντα που εισάγονται από την Ιαπωνία προ ευρωπαϊκέ χώρε. Τέλο πάντων, τα στοιχεία που είχαμε ω τώρα ήταν ικανοποιητικά. Ευχαριστούμε. Κυρία Λιωτά. Ευχαριστώ. Είναι πάντοτε δυσάρεστο να ακούει κανείς ότι μολύνονται, ρηπαίνονται νερό και τρόφιμα από ραδιενέργεια. Από τη ραδιενέργεια. Νομίζω ότι αυτό είναι πάντοτε κάτι που μας θλίβει. Θέλουμε να προστατεύσουμε λοιπόν τους πολίτες και την δημόσια υγεία. Οι επιστήμονες, πυρηνικοί επιστήμονες, έχουν ε, κάνει τις σχετικές μετρήσεις, γι' αυτό και εγώ έχω να θέσω ένα-δυο ερωτήματα προς την Επιτροπή. Προφανώς τα όρια για την περιεκτικότητα σαν διενέργεια των τροφίμων ε, έχουν ε, αναθεωρηθεί στην περίπτωση της Φουκουσίμα, έχουν μειωθεί. Είναι καλό αυτό και είναι θετικό στοιχείο για την ασφάλεια των τροφίμων. Χαμηλότερες τιμές προβλέπονται σε σύγκριση με το Δεκέμβριο. Μήπως έπρεπε λοιπόν να προβλέψουμε επίσημα όρια, διότι εάν στο όνομα της ασφάλειας των τροφίμων έχουμε συγκεκριμένα όρια, δεν ξέρω γιατί ξαφνικά αυτά μπορεί να αλλάζουν. Πώς μπορούμε να αλλάζουμε τα όρια για την Ιαπωνία και για άλλες χώρες. Ε, wird da später was zu sagen, was die θα μας πει ο κύριος Μίκος λίγο τι θα όριζε ως ε, χρονικό όριο για την ε, επιμόλυνση σήμερα την αργά. Κύριε Λεπάζ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα όσα είπε η κυρία Λιωτάρ, με δύο παρατηρήσεις επιπλέον. Η πρώτη έχει διαδικαστικό μάλλον ε, χαρακτήρα, γιατί όντως τίθεται το ζήτημα των προδιαγραφών. Άρα επιτροπολογία, άρα η ικανότητα που έχουμε εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωβουλευτέ να παρεμβαίνουμε όταν υπάρξει τροποποίηση των προδιαγραφών. Μα θέτουν πάντοτε ενώπιον τετελεσμένων ε, και πάνω απ' όλα διαπιστώνουμε την αδυναμία μα να αντιδράσουμε. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το διαπιστώνουμε, επανέρχεται διαρκώς το ίδιο πρόβλημα, επανεμφανίζεται και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εμείς ως εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης δεν μπορούμε να έχουμε λόγο για θέματα τόσο ευαίσθητα και σοβαρά για τον συμπολίτη μας. Είναι πολιτικό το ζήτημα μεν, αλλά, πάνω, αλλά πρέπει πιστεύω να επιμείνουμε ιδιαίτερος. Δεύτερο, επεσκέφθη την Ιαπωνία πριν από τρεις περίπου εβδομάδες, ένα μήνα, όπου στην περιοχή της ε, πόλης της Φουκουσίμα μπόρεσα να ε, καταγράψω την απόγνωση του πληθυσμού και την ε, κατάσταση ως προς τα διατροφικά ζητήματα και την ενημέρωση που τους προσφέρεται από τις αρχές για την ποιότητα αυτών των τροφίμων. Άρα πρέπει να επαγρυπνούμε πιστεύω και για τα επόμενα χρόνια, για τους επόμενους μήνες, γιατί ε, δεν είναι μόνο το κέζιο, είναι και το στρέζιο, είναι και πολλές άλλες ε, ε, ουσίες ραδιενεργές που πολλά αραμόρια ραδιενεργά που θα πρέπει να επαγρυπνούμε και που μπορεί να εμφανίζεται στα προστατοτρόφιμα για πολλά ακόμα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο, Μετά το Τσέρνομπιλ είδαμε ότι τα μανιτάρια και το θύραμα, το κρέας θυράματος εμφάνιζε τέτοια επιμόλυνση από ραδιενεργά. Δεν ε, υπάρχει δηλαδή ε, αυτόματη κατανάλωση ή εξαφάνιση αυτών των ραδιενεργών ε, από τη φύση. Παραμένουν και άρα παραμένει και ο κίνδυνος. Μισελ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως και η Κογίνα επισκέφθηκε και εγώ την Ιαπωνία. Έμεινα μια εβδομάδα εκεί, συζήτησα αρκετά με τους εκτροφείς ζώων, τους με τους όριζο καλλιεργητές και με τους πολίτες. Πρέπει να σας πω ότι ενημέρωση για τους πολίτες δεν υπάρχει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος εκεί τι σημαίνει ραδιενέργεια. Πρέπει να σας πω ότι ακόμη και εκεί που έγιναν οι ε, εθελοντικές λεγόμενες, εθελοντικοί λεγόμενοι εκτοπισμοί ή ε, και ε, χωριών, ο κόσμος εξακολουθεί να καταλώνει το ρίσκο που παράγει στο χωράφι του γιατί δεν έχει ιδέα για τη ραδιενέργεια και τον κίνδυνο που αυτή εκπροσωπεί. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους βουλευτές ότι στην Ιαπωνία δεν έχει ληφθεί υπόψη το ιστορικό του Τσέρνομπιλ. Δεν μοίρασαν παραδείγματι πλακέτες ιωδίου για να προστατευτούν τα παιδιά αλλά και οι ενήλικοι με το, από το πέρασμα του νέφους με το ραδιενεργό ιόδιο. Ενώ ξέρουμε ότι αυτό έχει γίνει και στο Κίεβο και στο Πρίτσιατ, οι Ρώσοι το κάνανε την εποχή του Τσέρνομπιλ, οι Ιάπωνες δεν το κάνανε. Για τα τρόφιμα. Και εδώ απευθύνομαι στην Επιτροπή και τη ζητώ να αναλάβει δράση. Διαρωτώ λοιπόν, ε, γιατί ε, διαρωτήθηκα τι κάνουν οι Ιάπωνες και πώ ορίζουν τα μέτρα του. Τι είχαν λοιπόν δείγματοληψία και μάλιστα πολύ περιορισμένη για να δούνε εάν πρόκειται κανεί να καταναλώσει ραδιενεργό γάλα. Άρα το σύστημα πολλέ πολλές φορές απεδείχθε ανεπαρκέ. Διότι διαπιστώθηκε ότι σε άλλε νομαρχίε υπήρχαν ε, υπερβάσεις των ορίων που είχαν οι ίδιοι Ιάπωνες ορίσει. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν μέτρα Υπάρχουν καλύτερα ενώσει πολιτών που κάνουν μετρήσει ε, στα τρόφιμα, γιατί πια ο κόσμο δεν έχει εμπιστοσύνη στι εθνικέ αρχέ Ιαπωνία. Α επανέλθουμε λοιπόν στην Ευρώπη τώρα. Είχαμε την έκθεση Μπελέ, η οποία προσδιορίσε προδιαγραφέ σε περίπτωση πυρηνική καταστροφή πυρηνικού ε, ατυχήματο στην Ευρώπη. Είχαμε στήσει από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τι προδιαγραφέ, γιατί είναι πολύ υψηλέ και τα παιδιά ιδιαίτερος έφταναν σε μερικούς μήνες μέσα να ξεπεράσουν τα αποδεκτά ετήσια όρια πρόσληψης φερρυπίν ραδιενεργού ιωδίου ή κεσίου. Θα ήθελα να επιθυμήσω ότι αυτές οι προδιαγραφές είναι πιο υψηλές από αυτές που έχουν ορίσει ως αποδεκτές οι ε, Ιάπωνες. Εμείς έχουμε 1000 μπεκερέλ, ενώ οι Ιάπωνες έχουν 500 μπεκερέλ ορίζει, ορίσει. Και γι' αυτό είχα απευθυνθεί στον κύριο Μπαρόσο και μάλιστα πρέπει να πω ότι η Επιτροπή δεν μας ενημέρωσε εγκαίρως. προσαρμοστήκαμε, ευθυγραμμιστήκαμε στις προδιαγραφές των Ιαπώνων. Παρακαλώ λοιπόν την Επιτροπή το είχαμε ζητήσει άλλωστε και με την έκθεση, να επανεξεταστούν αυτά τα επίπεδα με τις εκθέσεις Μπελέ σε περίπτωση έκθεσης κατά την ενέργεια. Και αυτό είπε και η κυρία Λεπά, πρέπει να εγγραφεί η συνθήκη τη Λισαβόνα, όχι στη συνθήκη Ευρατόμ, το μέτρο αυτό. Η δική τη συνθήκη βρατών είναι ούτω ή άλλω μεροληπτική, γιατί η δουλειά του είναι τα πυρηνικά. Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματο, οι ίδιοι για τη δουλειά του θέλουν να έχουν ε, υψηλότερα όρια ανοχή. Μου είπατε ότι από τους 800 τόσους ελέγχους είχαμε 8 ε, δείγματα που ξεπέρασαν πιο το όριο των 500 μπεκερέλ, έτσι. Μη μου λέτε λοιπόν, γιατί ε, το ορίζει το Ιαπωνικό, το επιμολυνσμένο με 200-300 μπεκερέλ στο κιλό, μην εννοείστε ότι αν καταναλώσει κανείς 200 μπεκερέλ, στο κιλο μην διανοειστε οτι αν καταναλωσει κανεις 200 μπεκερελ στο μπεκερελ το κιλό, μόνο και μόνο επειδή είναι κάτω από τα 500 το όριο, δεν κινδυνεύει η υγεία του. Εκπλήσουμε λοιπόν και χαστήσει από τον κύριο Μπαρόσο να μας πει ότι εντάξει έστω εισάγουμε πολύ λίγα προϊόντα από την Ιαπωνία, τσάι, κάποια σπανάκια κτλ. Γιατί να μην κάνουν αυτό που έκαναν και η Αυστραλία ή η Ινδία. Είπαν ότι δεν εισάγουν πια προϊόντα από την Ιαπωνία, αλλά προσφέρουν βοήθεια στην Ιαπωνία με άλλο τρόπο. Το να προσλαμβάνει κανείς ραδιενεργές ουσίες δεν σημαίνει ότι δεν διατρέχει κίνδυνο. Μπορεί να υπάρχουν στη φύση, αλλά είτε είναι το κέσιο το 34, είτε είναι το 37, το πλουτόνιο στα 30 χιλιόμετρα από το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα που εμφανίστηκε πρόσφατα, δεν αποτελούν κίνδυνο αυτά. Λοιπόν, το να μου λέτε ότι είναι πολύ λίγε οι εισαγωγέ, ε, δεν χρειάζεται παρά να σταματήσει η εισαγωγή των προϊόντων αυτών. Τσάι, σα αρέσει το τσάι. Ε, ναι, αλλά το τσάι αυτό παρουσιάζει 1500 μπεκέρε το κιλό ραδιενέργεια. Δεν είναι ανώδυνο αυτό, δεν είναι κίνδυνο. Άρα δεν πρέπει παρά απλώ να απαγορευτούν αυτέ οι εισαγωγέ. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρο. Κύριε Μίκο, ακούσατε τι ερωτήσει. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε αυτό που κάνουν και οι Αυστραλοί ποιες είναι οι τιμές οριακές, οι ανώτατες, οι κατώτερες, γιατί δεν, ακολου... γιατί δεν απαιτούμε τις χαμηλότερες οριακές τιμές από τους... και από τους Ιάπωνες. Γιατί δεν βελτιώνουμε την κατάσταση. Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Επιτρέψτε μου πρώτα να αρχίσω από το τέλος. Γιατί υποψιάζομαι ότι υπάρχει κάποια παρεξήγηση οτιδήποτε εξάγεται από τις εν λόγω νομαρχές της Ιαπωνίας ελέγχεται. Το 100% του, προσωπικού, του υλικού εξάγεται στην Ιαπωνία και επιπλέον αυτού γίνεται και επαλήθευση στην ευρωπαϊκή πλευρά σε δείγμα 10% στις εισαγωγές. Άρα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και γίνεται δύο φορές. Δεν είναι τυχαία δηλαδή η επαλήθευση που κάνουμε. Κάθε πράγμα που εξάγεται ελέγχεται. Εάν δεν ξεπερνά τα επίπεδα που έχουν προσδοριστεί στην Ιαπωνία δεν εξάγεται. Και γιατί εμφανίστηκε τότε ραδιενεργό τσάι στη Γαλλία και σε άλλες χώρες με 1500 μπεκέραλι το κιλό. Δεν αληθεύει αυτό που λέτε. Ναι, το ανέφερα και νωρίτερα στην ε, παρέμβασή μου. Ξεκινήσαμε με, τη, με την ε, νομαρχία της Φουκουσίμα και της ε, ζώνης απαγόρευσης αρχικά. Μετά επεκτείναμε όταν είδαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο πράσινο τσάι το μέτρο και στις λοιπές ε, νομαρχίες. Αντιδράσαμε όπως έπρεπε δηλαδή να αντιδράσουμε, γιατί δεν σταματάμε 100% τις ε, εισαγωγέ όπως η Αυστραλία και άλλες χώρες, γιατί θεωρούμε ότι θα ήταν δυσανάλογη η αντίδραση. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνο οι πληροφορίες ε, είναι υπό έλεγχο κάθε φορά και με το που θα εμφανιστεί το παραμικρό πρόβλημα αντιδρούμε. Δεν υπάρχει λόγος οι περιορισμοί αυτοί να καταστούν δυσανάλογα βαρύς για δε τα όρια. Προφανώς παρακολουθούμε τα ευρωπαϊκά όργανα, αυτά έχουν ζητηθεί. Δεν ήταν εύκολη καθόλου συζήτηση, αλλά υπάρχουν όρια. Μετά το Τσερνομπίλ ορίστηκαν τα όρια ως ασφαλή για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Γιατί μειώσαμε το όριο, τις τιμές μάλλον, απλούστατα διότι πρέπει να δείχνουμε συνέπεια ως προς την Ιαπωνική πλευρά. Γιατί τα εφιστάμενα επίπεδα στην Ιαπωνία, ανεξαρτήτως του λόγου, και δεν μπορώ να εκτιμήσω για ποιους λόγους και για ποιες λεπτομέρειες έχουν ε, ορίσει οι Ιάπωνες σε αυτό το επίπεδο. Επειδή είναι χαμηλότερο λοιπόν από το δικό μας, πρέπει και εμείς να δρούμε συντονισμένα από τη δική μας την πλευρά, άρα παρακολουθούμε τα επίπεδα που έχουν ορίσει οι Ιάπωνες, επειδή είναι χαμηλότερα από τα αποδεκτά στην Ευρώπη επίπεδα, που ήταν ήδη χαμηλά. Μηδενικός ο κίνδυνος, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς. Ήταν καλά βέβαια και τα ευρωπαϊκά όρια, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην συντονίσουμε τον έλεγχό μας σε αυτόν της ιαπωνικής πλευράς. <laughs> Μήπως ξέχασα κάποια ερώτηση? Καλώς. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά. Φυσικά θα συνοδεύσουμε, θα παρακολουθήσουμε, θα παρατηρήσουμε τις εξελίξεις τους επόμενους μήνες. Θα δούμε τι θα γίνει και θα συμβεί κατά τα τέλη του έτους, αν θα παραταθούν οι δοκιμές μέχρι το 2012. Και για τους Ιαπωνέζους ευχόμαστε ότι καλύτερο για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το τρομακτικό ατύχημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν σημαντικό να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση σίγουρα. Και συνεχίζουμε τώρα αμέσως με το σημείο που είχαμε ξεχάσει και είχαμε αφήσει εχθές, το 17, σημείο 17. Προφορική ερώτηση <clears throat> σε σχέση με τις ε, επιπτώσεις των διαταρακτών ενδοκρινικής λειτουργίας. Ε, είναι ε, παρούσα. Θα ζητούσα από πλευρά και του Πάτρικ Μόρβι από πλευρά τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσουν αυτή την ερώτηση. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ, να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Μια σύντομη επισκόπηση θέλω να σας παρουσιάσω για το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους διαταρακτές που είναι ένα σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρησιμοποίησαμε την τέταρτη εφαρμοστική έκθεση φέτος τον Αύγουστο βάσει της ανακοίνωσής μας για τους ενδοκρινικούς ταράκτες και εκεί ε, αναφέραμε όλα τα τελευταία βήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με την έρευνα, την αύξηση των ε, τραπεζών δεδομένων που έχουμε και των σχετικών πληροφοριών, την άντληση πληροφοριών από, τη, από το ΡΙΤ, τις σχετικούς κανονισμούς της Επιτροπής, ισχύοντας και μελλοντικού. Η στρατηγική που έχει καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον κάπως παλιά, από το 1999. Μετά από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου είχε υιοθετηθεί τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται κατά πόσο μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση αυτής της στρατηγικής καθώς και νέα κριτήρια εντοπισμού των ε, διαταρακτών. Ίσως και βάσει του νέου κανονισμού για το ΡΙΤΣ και μιας νέας επιστημονικής θεώρησης πια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Επειδή η στρατηγική μας λοιπόν ανάγεται στο 99 και επειδή έχουμε πολλές ρυθμιστικές υποχρεώσεις, ξεκινήσαμε μια ευρεία μελέτη για να δούμε τι επιστημονικά στοιχεία διαθέτουμε για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, καθώς και τις δυνατότητες ή τα επιστημονικά κριτήρια που μπορεί να ισχύουν πλέον για τον εντοπισμό των ουσιών αυτών. Η μελέτη θα είναι έτοιμη στα τέλη της χρονιάς και θα δημοσιευτεί βάσει των πορισμάτων της επίσης. Θα υπάρξουν ανταλλαγές με ενδιαφερομένους, καθώς ε, σκοπεύουμε να οργανώσουμε μια σημαντική διάσκεψη κατά τη διάρκεια του 12 για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Εδώ έχουμε αρκετέ δυνατότητε. Πρώτα απ' όλα να αναθεωρήσουμε και ίσω και να ανασυστήσουμε την ισχύουσα ευρωπαϊκή στρατηγική και έπειτα να ανταποκριθούμε στι ρυθμιστικέ υποχρεώσει. Στου κανονισμού για συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να εξεύρουμε και ανάλογα κριτήρια μέχρι το 2013 αλλά και θα πρέπει να δούμε πάλι το τι ισχύει για τους διαταράκτες ε, στα πλαίσια του REIT ε, και αυτό να έχει ολοκληρωθεί ως διαδικασία το 2013. Στενά επίσης παρακολουθούμε τι συμβαίνει στον ΟΣΑ και στον ΠΟΕ. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για τους ανθρωπινικούς διαταράκτες και συνειδητοποιούμε ότι όχι μόνο συσσωρεύονται στοιχεία για το θέμα αυτό, αλλά και περισσότερε ανησυχίες. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μείγματα. Το 2009 η Επιτροπή ξεκίνησε μία σοβαρή μελέτη με θέμα την τοξικότητα σε συνδυασμού και μείγματα ουσιών. Τα απορίσματα της έκθεσης αυτής διατέθηκαν τον Φεβρουάριο του 2010 και μετά τη δημοσίευσή του διοργανώσαμε διάφορους γύρους συνομιλιών με με τους ενδιαφερομένους, μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Οπότε στην αρχή της φετινής χρονιάς ζητήσαμε και επίσημη γνωμάτευση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία και το Περιβάλλον. Το αίτημά μας υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο. Ελπίζουμε να έχουμε επιστημονική τοποθέτηση τη Επιτροπή το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο. Βάσει τη συνεισφορά αυτή και όλο το άλλο που θα συγκεντρώσουμε θα καταρτήσουμε έκθεση για το πώ οι συνδυασμοί ουσιών μπορεί να επηρεάζονται από το... ή να επηρεάζουν και το νομοθετικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα και ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εξετάζει μεμονωμένα τις χημικές ουσίες και από την χημική μόνον άποψη. Ίσως πρέπει πλέον να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με τα μείγματα χημικών ουσιών. Με 100.000 χημικές ουσίες ε, στα παρατήματά μας, οι δυνατότητα συνδυασμού είναι πλέον άπειρες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι επιστημονική πείρα διαθέτουμε και τι επιστημονικά στοιχεία για τα μείγματα αυτά που μπορεί να αποτελούν ε, πραγματικό κίνδυνο για τον ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Κυρία Μακέβαν. Θα θέλω να ευχαριστώ την Επιτροπή για την ενημέρωση. Χαίρομαι που υπάρχει κάποια δραστηριοποίηση. Έχουμε πει ότι το θέμα αυτό είναι παλιό. Θέλαμε να δούμε τι γίνεται με τις ουσίες των ενδοκρινικής λειτουργίας και τις επιδράσεις κοκτέιλ. Ξέρουμε ποιε είναι, υπάρχουν κατάλογοι των ουσιών αυτών. Πλέον επίγει να αναλάβουμε δράση. Και νομίζω ότι υπάρχει και εξέλιξη από πλευρά των Η Γερμανία προσέθεσε πρόσφατα κάποια ουσία στον κατάλογο. Άρα πρέπει να δράσουμε, επίγει. Δεν αρκεί πια να μιλάμε μόνο. Και βεβαίως καταλαβαίνω ότι στην αξιολόγηση των ε, ουσιών διατάραξης ενδοκρινικής λειτουργίας. Υπάρχουν διαφορετικές ε, ε, προσεγγίσεις μεταξύ Γερμανίας και Δανίας, Φερρυπίνη. μία έχει την προσέγγιση του κινδύνου και η άλλη της διακινδύνευσης. Πώς το αντιμετωπίζετε σε αυτό, πώς το βλέπετε. Μια δε μη κυβερνητική οργάνωση μου λέει ότι στον κανονισμό περί ζυζανιοκτώνου του προηγούμενου, από τον Ιούνιο του 2011, προβλέπεται ότι δεν μπορούμε να εγκρίνουμε ουσία που ε, θεωρείται ότι έχει ε, σαν συνέπεια τη διατάξη ενδοκρινικής λειτουργίας, συνέπεια στην υγεία. Αλλά τον Σεπτέμβριο, λέει, τον προηγούμενο μήνα δηλαδή μόλις, ένα προϊόν Procloaz ε, το όνομα, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς αξιολόγηση των ε, ιδιωτήτων του, των σχετικών με τη διατάρξη ενδοκρινικής ε, λειτουργίας, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν ε, από τη σχετική φιλολογία διαπιστωμένες συνέπειες στην ενδοκρινική λειτουργία και το BioFairfin επίσης που θα έχετε να συστήσετε στο μέλλον φαίνεται που παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα. Εσείς μιλάτε για το τέλος του 2013 στο χρόνο διάγραμμά σας, ενώ τα κράτη-μέλη ήδη θα έπρεπε να αποκλείουν την αδειοδότηση τέτοιων ουσιών. Σχολιάστε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Μαγκάβαν. Κρίσταλ Σόλτιμος. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να συμμετάσχω στη συζήτηση της Επιτροπής σας και δεν είμαι μέλος τακτικό αλλά της ύμκο. Ευχαριστώ πολύ για τις, ερωτήσεις της, ε, για τις απαντήσεις ερωτήσεις μας και αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή ε, το επεξεργάζει το θέμα αυτό, όπως είπε και η Λίνδα. Δεν μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία για να είμαι πιο ευθεία στην ερώτησή μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα γιατί πρέπει κάτι να γίνει. Όπως θα γνωρίζετε ίσως η Προεδρία της Δανίας που ξεκινάει στο πρώτο εξάμεινο του 2012 στις προτεραιότητες της για τη δημόσια υγεία έχει ακριβώς την αντιμετώπιση των, του προβλήματος των ουσιών που διαταράσσουν την κλινική λειτουργία. Η δε καινούρια κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει απαγόρευση αυτών των ουσιών, ιδιαίτερων, ιδιαίτερος εκείνων που θεωρούνται πιο επικίνδυνες, πολύ επικίνδυνες. Δηλαδή έχουν μάλλον μια ε, προληπτική προσέγγιση στην νομοθεσία για να προστατευτεί η δημόσια υγεία, η υγεία του καταναλωτή. Αυτό μπορείτε να το σχολιάσετε. Είναι κάτι το οποίο βλέπετε και εσείς σαν δυνατότητα για το μέλλον προς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Βέστλουντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω μια-δύο ερωτήσει γενικότερου χαρακτήρα. Γιατί πρόκειται για ένα πρόβλημα ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ταυτόχρονα όμω διαπιστώνουμε ότι έχουμε πρόβλημα και στην νομοθεσία μας γιατί θα έπρεπε μάλλον όλα τα ζητήματα αυτών των ουσιών ε, να τα εξετάζουμε ως πρόβλημα που προξενεί κάθε ουσία χωριστά, μεν, αλλά να κοιτάμε και τα κοκτέιλ, δηλαδή τη συνεργατική σχέση μεταξύ των ουσιών. Επίσης θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ε, κοινοποιούν πληροφορίες που ενδεχομένω έχουν ε, για τις ουσίες αυτές. Πολύ καλά, ισχύει η αρχή και δεν είναι κακή. Αλλά ε, από την άλλη αν υπάρχει κάποια έρευνα, αποτελέσματα έρευνας ε, για την υπόθεση αυτή, δεν θα πρέπει και αυτή να κοινοποιείται και αν ε, διαπιστώνετε ότι οι επιχειρήσει Φερπίν δεν κάνουν την έρευνα που θα έπρεπε. Ποιο φέρει την ευθύνη. Πώς θα ελεγχθεί ότι είναι καλά τα στοιχεία που έχουμε, ότι υπάρχει επαρκή έλεγχο, αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα το βλέπουμε και στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές, στα χημικά. Πρέπει να έχουμε πιο αξιόπιστη έρευνα. Πρέπει να εστιάσουμε την έρευνά μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στους παράγοντες αυτούς κινδύνου και ανησυχίας. Τι θέλει, επομένως, διαφορετικά το ζήτημα ε, ως προς τις επιπτώσεις χαμηλών δόσεων ή κάποιων άλλων ουσιών που ενδεχομένως δεν καταγράφονται στην νομοθεσία. Δεν πρέπει να γίνει η σχετική προσπάθεια έρευνας ε, από τις αρχές. Και έχω ακόμη μια ερώτηση στα όσα υπόθηκαν νωρίτερα το ριτς είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Αλλά ο καταναλωτής το βρίσκει πολλές φορές ε, ε, εμπόδιο διότι υπάρχουν χημικές ουσίες που είναι γνωστό ότι προξενούν κίνδυνο αλλά δεν έχουν επαρκώς καλυφθεί και πάνω απ' όλα δεν έχουν εξασφανιστεί επαρκείς εναλλακτικές η μπισφενόλη φερρυπίνη, άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις κονσέρβες ή που ενδεχομένως να αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την έγκυο γυναίκα. Είναι λοιπόν το πρόβλημα γενικότερο. Δεν θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί και αυστηροί στα προϊόντα που καταναλύσκουμε, δεν θα έπρεπε να ακολουθούμε και την αρχή της υποκατάστασης όταν υπάρχει μια εναλλακτική υγιή σε κάποιο προϊόν, δεν θα πρέπει να την προωθούμε πάντα. Η Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο στον Κρήτονα Αρσένη, θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα σε αυτό που υπόθηκε για την πισφενόλη Α. Η ΆΣΕΣ που είναι η Γαλλική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων δημοσίευσε δύο εκθέσεις για, την, για τους κινδύνους για την υγεία της Μπισφενόλης Α με αποδεδειγμένα για το ζώο και υπο, ύποπτα για τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο ε, συνέπειες στην δημόσια υγεία και ρωτώ ποια είναι η κατάσταση. Έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις, 2006-2007, δεν έχουν αναθεωρηθεί, δεν έχουν ανατραπεί. Γιατί περιμένουμε, γιατί δεν αναλαμβάνουμε δράση. Όταν έχουμε να κάνουμε προϊόν με τεράστιες συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου, οικονομικές επίσης, όχι μόνο ε, κοινωνικές αλλά και οικονομικές, γιατί βέβαια πληρώνει το κοινωνικό ταμείο την... Ε, ε, την κάλυψη του ανθρώπου που βρίσκεται στο νοσοκομείο που είναι άρρωστος, γιατί να μην είμαστε πολύ πιο ε, αποφασιστικοί στη δράση μας, γιατί να μην προλαμβάνουμε, γιατί να μην είμαστε προμηθείς ο Κρήτον. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη μελέτη του Γαλλικού Ιδρύματος που λέει ότι αποδεικνύονται οι συνέπειε αυτές, οι επιπτώσει και στην ανθρώπινη και τη ζωική υγεία. Εντοπίζει ευάλωτου πληθυσμού, παιδιά, νεογνά, έγκυου γυναίκες και ζητά την αντικατάσταση σε όλα τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Αναφέρεται επίσης ότι οι επιπτώσεις εντοπίζονται και σε δοσολογίες πολύ χαμηλότερε από τα γνωστά και τα επιτρεπόμενα όρια. Είναι λοιπόν πολύ περίεργο το πρόγραμμα της Επιτροπής, όπου τον Ιούνιο του 2013 η Επιτροπή θα αναθεωρήσει αν κάποιες ουσίες που ε, διαταράσουν ενδοκρινικά την ε, ανθρώπινη υγεία μπορεί να ε, περιληφθούν σε κατάλογο και να αλλάξουν τα ωριά τους. Εάν λοιπόν υπάρχει ασφαλής εναλλακτική, η Επιτροπή απλώς θα αποφασίσει εάν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες θα αντικατασταθούν με άλλους. Και όλα αυτά από το 2013. Ενώ ήδη είναι συντριπτικά τα επιστημονικά στοιχεία. Έχουμε πλέον δεδομένα για τις επιπτώσεις. Είναι οι θαλίτες, και άλλες τόσες ουσίες. Γιατί να χρησιμοποιούμε λοιπόν τέτοια υλικά. Ακόμη και αν δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτή τη στιγμή την τεσθενόλη α στα πλαστικά σκεύη, ίσως να μην είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις. Νομίζω λοιπόν η Επιτροπή για αυτό το τόσο επίγον ζήτημα χρονοτριβεί ιδιαίτερος είναι καθοριστική σημασία για τη δημόσια υγεία. Και εγώ ίδιο, και από ό,τι κατάλαβα και πολλοί άλλοι συνάδελφοι θα σας παρακολουθούμε στενά. Σας παροτρύνουμε λοιπόν να μας υποβάλλετε κάποια πιο συγκεκριμένη πρόταση και συντομότερα. Ε. Ευχαριστούμε. Ο Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές όταν ε, αναφέρονται στο πόσο κατεπήγον είναι το ζήτημα. Και εμείς στις παρατηρήσεις μας δεν πάβουμε να το λέμε ότι θεωρούμε το θέμα αυτό επίγον. Και κάποια άλλα στοιχεία ήθελα να αναφέρω και εκ μέρους της κυρίας Παρφανόβα, να το πω και αυτό πριν το ξεχάσω βλέπουμε οι ενδοκρινικοί διαταράκτες να περιλαμβάνονται σε πάρα πολλά προϊόντα που έρχονται στα χέρια των καταναλωτών, σχεδόν στα πάντα. Άρα είναι πολύ υψηλό ο κίνδυνος για την βιομηχανία την ίδια και πάνω απ' όλα για την ανθρώπινη υγεία. Το ερώτημά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι η Γενική Διεύθυνση είναι επιφορτισμένη με θέματα υγείας το εξετάζει αυτό. Υπάρχει προβληματισμός εντό επιτροπή για το θέμα αυτό, εφόσον είναι τόσο υψηλά τα διακυβεύματα και μας ανησυχεί τόσο πολύ το θέμα αυτό. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι το ίδιο. Πώς πιστεύετε ότι ο βιομηχανικό αυτός κλάδος μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτή την συζήτηση. Μπορεί να κινηθεί προς την κατάργηση αυτών των ενδοκρινικών ε, διαταρακτών σύντομα. Πληροφορίες, ερευνητικά στοιχεία διατίθενται. Πολεμάμε όλοι στο ίδιο στατόπεδο για τον ίδιο σκοπό, την ανθρώπινη υγεία ή υπάρχουν ισχυρές πιέσεις μεταξύ των πολιτικών ηθινόντων και των βιομηχανικών υπευθύνων που μπορεί να παρακολουθήσουν τις προσπάθειές μας να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Merci. Ευχαριστούμε. Ο Σλούτερ παρακαλώ. Ευχαριστώ τους αρμόδιους για αυτή τη συζήτηση από πλευρά τη επιτροπή μα. Ε, και εγώ πιστεύω ότι η ενδοκρινική διαταράκτηση είναι μία από τι πιο υποτιμημένε απειλέ έναντι ε, της ανθρωπότητας που αντιμετωπίζουμε και η έκθεση σε αυτά όταν είναι κανείς ε, νεογνώ ή μωρό μπορεί να είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη και είναι εκπληκτικό ότι βλέπουμε αυτές τις ουσίες ε, εσκεμμένα να προστίθενται σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε στην επιδερμίδα μας ε, και ε, που έχουν σε επαφή και χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, σε κάψιμα, στις εξατμίσεις των οχημάτων, στα ρούχα, σε πάσης φύσεως προϊόντα χρησιμοποιούνται αυτές οι χημικές ουσίες και έρχονται σε επαφή με το σώμα μας ή παντού που ζούμε και στην, ε, στον καθαρισμό ρούχων και τα λοιπά. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό το ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το μεγάλο κίνδυνο και δεν εγγράφονται αυτές οι ουσίες ε, στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών σε σχέση με την μελέτη χημικών προϊόντων έγινε μια εξέταση εκατοντάδων τέτοιων χημικών ουσιών που έχουν διαταρακτική επίπτωση και επελέγει σε σχέση με ε, τις ε, ιδιότητες ε, επελέγησαν οι ουσίες αυτές διότι στο REACH υπάρχει μεγάλη, μεγάλος κίνδυνος δεν είναι, όλοι δεν είναι όλες πρωτογενείς ουσίες, ε, βρίσκονται, έχουν κάποιες, ε, ε, κάποιες ιδιότητες διαταράκτη, αλλά δεν έχουν ε, εγγραφεί σε αυτόν τον κατάλογο. Για παράδειγμα όσον αφορά την τοξικότητα, αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση αυτή τη μελέτη που είναι εξαιρετική μετά από τις 319 αυτές ουσίες εξετάστηκε σε, βά σε βάθος ε, ποιες από αυτές τις ουσίες ε, θα εντασσόντουσαν στα πλαίσια του ριτς ε, και ποιες θα εντασσόντουσαν ή όχι και υπήρξαν και κάποιες εξαιρέσεις μετά εξετάστηκαν άλλες χρήσεις με βάση το ριτς κατέληξαν λοιπόν στην πρόταση για 22 αποδεδειγμένες τέτοιες ουσίες που έχουν τέτοια διαταρακτική επίπτωση και Ας ξεκινήσουμε με αυτές τις 22 ουσίες ε, σε αυτό τον ε, κατάλογο, διότι αυτές είναι οι χημικές ουσίες για τις οποίες κάνω ακριβώς λόγο. Είναι οι φθαλικές ουσίες που έχουμε σε πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, τα φθαλικά, οι ε, καμφορές και οι διάφορες ενώσεις που χρησιμοποιούμε στην επιδερμίδα μας. Έχουμε τις προσθετικές ουσίες καυσίμων ε, οχημάτων. Αυτές είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με αυτές και ξέρουμε ότι έχουν διαταρακτική επίπτωση ενδικρονολογικά γιατί να μην δούμε αυτούς τους 22 φακέλους και να ζητήσουμε από την υπηρεσία, από την οργάνωση να εγγραφούν στον απαγορευμένο κατάλογο. Αν δεν γίνει αυτό θα έχουμε τεράστιες επιπτώσεις βάρος της υγείας και δεν θα καταφέρουμε να ε, καταλήξουμε σε μια δράση που να προστατεύει την υγεία. Αυτές οι 22 ουσίες θα ήταν εξαιρετικές για να εγγραφούν σε αυτόν τον κατάλογο. Θα παρακαλούσα να προετοιμαστούν αυτά τα χαρτοφυλάκια προς περαιτέρω ε, επεξεργασία και να βοηθήσουμε έτσι για την προστασία της κοινωνίας και της υγείας μας και να βρούμε και εναλλακτικέ ουσίες για να αντικαταστήσουν αυτές ε, όταν θα απαγορευτούν. Θα ήθελα να ζητήσω να εγγραφούν σε αυτόν τον κατάλογο. Έχουμε μια στρατηγική για 12 έτη. Τι γίνεται σε σχέση με τις δράσεις μας. Θα μπορούσε αυτή να είναι η πρώτη συγκεκριμένη χειροπιαστή δράση από τη σκόνη στα δωμάτια των παιδιών μας Πού βρίσκεται το υψηλότερο επίπεδο φθαλικών ουσιών, στη σκόνη και στα υπνοδωμάτια των παιδιών μας. Μπουσουλάνε στο πάτωμα και εισπνέουν αυτές τις ουσίες. Απόλυτα απαράδεκτο. Γκερμπράντι, έχεις δίκιο. Οι βιομηχανικοί κύκλοι τροχοπεδούν τις εξελίξεις. Θα ήθελα όμω ε, σε σχέση με τι ουσίε αυτέ να βρίσκονται εκτό των υπνοδωματίων των παιδιών μου και δεν είμαι ο μόνο που έχει αυτό το αίτημα και σίγουρα υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν. Λοιπόν, σας παρακαλώ, εξετάστε την πρότασή μου. Αυτές οι 22 ουσίε να ενταχθούν στον κατάλογο υποψήφιων υπό απαγόρευση ουσιών. Ε, και θα ήθελα να προτείνω για τα κοκτέιλ, για τα μείγματα αυτών των χημικών. Όλοι είμαστε εκτεθειμένοι σε, αυτές τις, ε, σε αυτά τα μείγματα ουσιών και πρέπει να κάνουμε κάτι εναντίον αυτή τη κατάσταση. Και εγώ μπορώ να προσθέσω την φωνή μου άρρηκτα σε αυτά. Κάνουμε λόγο για αυτά τα θέματα και την έχουμε και στην οδηγία για την προστασία των φυτών στη Γεωργία. Τα ξανασυζητήσαμε πάλι και όταν έχουμε τα θέματα βιοκτώνων. Και η ερώτησή μου είναι προς τον κύριο Μέρφυ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξεκινάμε με ένα υπερβολικά μεγάλο εύρος όταν συμπεριλαμβάνουμε αυτά τα μείγματα, αυτά τα κόκτέιλ. Θέλουμε να τα γνωρίζουμε όλα και στο τέλος τέλος δεν θα ήταν πιο σωστό να έχουμε ένα στενότερο πλαίσιο, να επικεντρωθούμε σε ένα στενότερο κύκλο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Όταν έχουμε ένα τεράστιο εύρος φάσματος και όλες, όλα τα ενδεχόμενα θέλουμε άμεσα να τα καλύψουμε, ίσως ε, ζητάμε κάτι υπερβολικό σε σχέση με τα όσα μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ακριβώς όσον αφορά τους ενδοκρινολογικούς, ενδοκρινικούς διαταράκτες έχουμε και το σημαντικό τμήμα των ιατρικών προϊόντων που δεν το έχουμε θέσει στο επίκεντρο. Εκεί όμως βρίσκονται πάρα πολλά φλέγοντα θέματα τι είναι αυτά τα οποία καταλήγουν στο νερό, στους υδάτινους πόρους και παραμένουν επί δεκαετίες εκεί, στο, στα νερά, στο υπέδαφος, στον υδάτινο ορίζοντα. Και συζητώντας για την οδηγία, για την προστασία των υδάτινων πόρων, αυτά πρέπει να τα δούμε. Και θα έπρεπε να κινητοποιηθούμε. Θα επιθυμούσε ο κύριος Μέρφυ να μας πει κάτι. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να έχουμε μια λογική, ένα λογικό αποτέλεσμα με βάση αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστώ. Sophie Oconi. Ευχαριστώ, Σοφία Κονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν. Συμφωνώ απολύτω. Όλοι γνωρίζουμε τι συνεπάγεται το ζήτημα αυτό προ τη δημόσια υγεία. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα που χρειάζεται. Και θα συμφωνήσω με την κυρία Κλάση εδώ. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να δει κανεί την κατάσταση. Υπάρχουν τα στοιχεία που έχουμε, δεδομένα που γνωρίζουμε για ορισμένα προϊόντα και αυτά στα οποία θα πρέπει να κάνουμε κάποιε επιλογέ. Για τι φενόλε, τι θανάλατε, τη βιοφενόλη, τη βιφενόλη, διορθώνω μου λέτε α, ε, που γνωρίζουμε ότι είναι επικίνδυνα, που ξέρουμε ότι έχουν συμμετοχή ή συμπεριλαμβάνονται, εν πάση περιπτώσει, στον τρόπο προσδορισμού ε, συντήρησης ε, των τροφίμων και έχουν συνέπειες. Ξέρουμε ότι παραδείγματι υπάρχουν ουσίε που εμφανίζονται όταν κάποιο προϊόν το ξαναθερμαίνει ο καταναλωτή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον υποχρεωτική σήμανση της ύπαρξη ενό τέτοιου προϊόντος ε, στην ε, συσκευασία έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι υπάρχει κίνδυνος μετάλλαξη στην ώρα που θερμαίνει το προϊόν στα τρόφιμα. Δεν πρέπει να γίνει σχετική ενημέρωση πρώτα απ' όλα στον καταναλωτή για να του εξηγήσουμε. Γιατί περιμένουμε ε, για να... Ε, ε, περιμένουμε βέβαια να λαμβάνεται η σχετική νομοθεσία και τα μέτρα κτλ. Αλλά πέραν αυτού που συμφωνώ ασφαλώς δεν θα έπρεπε να βάζουμε και σαφή σήμανση πάνω στα προϊόντα και με τον τρόπο αυτόν να προ ειδοποιούμε τον καταναλωτή και να του ζητούμε να φροντίζει να παίρνει και εκείνο στα μέτρα του για τη χρήση ορισμένων τροφίμων. Αυτά. Ευχαριστώ. Έχουν καλυφθεί τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέρφυ. Άλλες παρεμβάσεις όχι κύριε Μέρφυ. Πρόεδρε, θα ήθελα εσείς να με καθοδηγήσετε λίγο πόσο χρόνο έχω για να απαντήσω. Έχετε πέντε λεπτά, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώ λοιπόν, θα αναφερθώ στις ε, κατά παρατηρήσεις των βουλευτών, που να τις καλύψω όλες. Ως προς τον εντοπισμό των ε, ουσιών για τα ενδοκρινικής λειτουργίας. Ένα από το πρόβλημα τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι πολλά είναι τα χημικά που έχουν συνέπεια και επίπτωση στο ενδοκρινικό σύστημα, όπως ο καφές περίπου. Πολλά από, τα, από τις ουσίες που καταναλώνουμε καθημερινά, δηλαδή, επηρεάζουν την ενδοκρινική λειτουργία. Το θέμα είναι πότε είναι ε, δυσμενής αυτή η διατάραξη και οι επιπτώσεις μπορούν να σημαίνουν ακόμη και κίνδυνο για το για την επιβίωση του είδους, εάν πιστέψουμε τις ε, μετρήσεις των δανών ε, ως προς ε, την πυκνότητα του σπέρματος της χώρας της Βόρειας Ευρώπης, υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για την επιβίωση του είδους. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε εάν υπάρχει επίπτωση κατά πόσο αυτή είναι δυσμενής και κατά πόσο μπορούμε τις επιστημονικές, τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε να τα μετατρέψουμε σε ε, κάποια συνέπεια, να τα αξιοποιήσουμε δηλαδή. Και θα ήθελα να πω ότι ναι, υπάρχει νομοθεσία, εφαρμόζεται ο κανονισμό και ενώ περιμένουμε την εξέλιξη των προτάσεων τη ευρωπαϊκή Επιτροπή για κριτήρια εντοπισμού των ουσιών για τα εξεδοκρινικές λειτουργία, υπάρχουν κατά πρωτογενή κριτήρια θα έλεγα, που εφαρμόζει ο κανονισμό, που ορίζει ο κανονισμό και που λέμε ότι αν ταξινομείται με βάση κάποια κριτήρια μια ουσία, με βάση την ταξινό, ταξινόμηση, τότε θεωρείται ότι είναι ουσία διατάραξη ενδοκρινική λειτουργία και άρα εφαρμόζεται αυτό ο περιορισμό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 απαιτείται να καταθέσει προτάσει για τα για κριτήρια που θα αντικαταστήσουν τα προσωρινά κριτήρια. Άρα εφαρμόζεται ο κανονισμός και έτσι η Επιτροπή έχει περισσότερο ε, διάστημα ακόμη στη θέση της για να εισαγάγει τις μόνιμες ε, διατάξεις. Με δύο χρόνια ακόμη δηλαδή. Επίσης, επιτάχυση των ε, διαδικασιών. Να σας πω, είναι μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ζήτησε από τον αντισυμβαλόμενο να διαθέσει όλες τις πιστάμενες πληροφορίες ως προς τα επιστημονικά δεδομένα που, οδηγούν. που ως προς τις ε, συνέπειες αυτών των ουσιών διατάραξης δοκρινικής λειτουργίας μας έδωσε χιλιάδες σελίδες μελετών που αφορούν αυτέ τι ουσίε Και ναι, μεν υπάρχουν κάποιε θέσει που λένε ότι κάποιε ουσίε είναι ουσίε διατάραξη ενδοκρινικής λειτουργία. Στη συζήτηση όμω που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με επιστημονικού συνεργάτε επιρρογνώμονε κτλ. και όπου ρωτήσαμε συγκεκριμένα τι είναι, ποια ουσία είναι ε, διαταράξη στην ενδοκρινική λειτουργία, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουν μεταξύ του επιστήμονε. Όπως είπα, η έννοια του συνδυασμού ή του κοκτέιλ ε, ακόμη δεν έχουμε βάση για λήψη αποφάσεων. Και γι' αυτό στρεφόμαστε προς επιστημονικές επιτροπές, Επιστημονική Επιτροπή Υγείας και Περιβάλλοντος Φερρυπίν και διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας και για το συνδυασμό, δηλαδή για το κοκτέιλ, για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει και με βάση αυτά που θα μας πούνε προσπαθούμε και εμείς να λάβουμε τις αποφάσεις μας με βάση βέβαια τα επιστημονικά δεδομένα στο βαθμό που μπορούμε. Έτσι λοιπόν, για την ΑΝΣΕΣ και την Πισφενόλη Α που ανέφεραν πολλοί ομιλητέ. Έχει εκδώσει και η ΕΦΣΑ μια γνωμοδότηση πριν από ένα-δύο χρόνια για την Πισφενόλη Α και τη χρήση της ε, σε μπιμπερών και σε δοχεία που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Στα μπιμπερών λοιπόν έχουμε τώρα δεδομένη την έκθεση ANSES και θα ζητήσει η υπηρεσία μας από τη ΣΑΝΚΟ δηλαδή να αξιολογηθεί η έκθεση της ΑΝΣΕΣ από την ΕΦΣΑ και να δούμε αν υπάρχουν νέα στοιχεία σε σχέση με την έκθεση ΆΝΣΕΣ και να δούμε αναλόγω αν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι στις νομοθεσίες, στη θέση μας, στη στάση μας απέναντι σε αυτά. Είμαστε ενήμεροι πάντως για την έκθεση ΆΝΣΕΣ. Και καθώς η ΕΦΣΑ έχει την ευθύνη για την ε, γνωμοδότηση αυτή, του ζητούμε, θεωρούμε ότι το του είναι αυτό. Δηλαδή, ζητήσουμε από την ΕΦΣΑ να αναθεωρήσει, εάν το θεωρεί σκόπιμο, την γνωμοδότηση αυτή. Τώρα, για το αν υπάρχει παρέμβαση ή στήριξη από την ε, βιομηχανία. Ασφαλώς θα συμφωνείτε ότι σε κάθε θέμα υπάρχουν ε, αντικρουόμενες απόψεις, το μεν και το δε υπάρχει χρησιμότητα να συζητούνται όλα τα ζητήματα. Και αυτό μπορεί να κάνει η Επιτροπή μόνο είναι να ακολουθήσει μια αντικειμενική γραμμή με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Αυτό προσπαθούμε να πράξουμε. Για τι επιπτώσει των συνδυασμών ουσιών, το κοκτέιλ δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο πιθανό αριθμό συνδυασμών ε, ουσιών που ε, βρίσκονται στο περιβάλλον είναι τεράστιος Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να εντοπίσουμε επακριβώς το συνδυασμό εκείνων που θεωρούμε κατά προτεραιότητα να μελετήσουμε. Άρα αυτό που θέλουμε πρώτα απ' όλα είναι να κάνουμε με βάση τα δεδομένα της παρατήρησης μια προεπιλογή για το σε τι μπορεί να εκτίθεται ο πολίτης ε, περισσότερο, κατά πλειονότητα. Πριν από δύο χρόνια η Δανία έκαναν μία μελέτη με βάση την έκθεση παιδιών 18 μηνών ε, και τις συνέπειες στην ενδοκρινική λειτουργία από τα πλαστικά μπιμπερών που χρησιμοποιούνταν και μας ε, κάλεσαν να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό μέσω της νομοθεσίας. Είναι μεγάλη πρόκληση όμως. Γιατί πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο τις μεμονωμένες ουσίες, αλλά συνδυασμούς ε, σε 7, 8, 9 διαφορετικά νομοθετικά κείμενα και ταυτόχρονα εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των κοκτέιλ αυτών των ε, σύνθετων ουσιών δηλαδή, πρέπει να λάβουμε υπόψη και να προσαρμόσουμε αναλόγως νομοθεσία που βρίσκεται σε διαφορετικά επίπεδα. Και αυτό πρέπει να γίνει κατά τρόπο βέβαια οικονομικό και αποτελεσματικό για να μην πετάμε τα λεπτά μας από το παράθυρο. Η, ουσία των 20, η λίστα των 22 ουσιών που έχει εντοπίσει η Κέμψε και παραδείγματι έχουμε και για το αν θα πρέπει αυτές να ε, παγώντα το REACH. Δεν μπορώ να σα δώσω κάποια, κάποια εγγύηση τώρα ότι θα μπουν στον κατάλογο αυτών. Ξέρω ότι κάποια κράτη-μέλη θα, θα παρακολουθήσουν την κατάσταση και θα ετοιμάσουν προτάσει για το παράρτημα 15 για να ενταχθούν αυτέ τι ουσίε στη διαδικασία του REACH. Από την άλλη βεβαίω υπάρχει ανταγωνισμός, ότι θα πρέπει να μπει σε αυτόν τον κατάλογο και διαφωνία ε, για τις ουσίες διατάραξης της ενδοκρινικής λειτουργίας. Ε, θα πρέπει να δούμε αν αυτό έχει να κάνει συγκεκριμένα με την αναπαραγωγική λειτουργία ή κάποιες άλλες συνέπειες στον οργανισμό και αναλόγως της ε, επιλογής στη συνέπεια θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ουσίες που μελετάμε κατά προτεραιότητα. Άρα το φιλτράρισμα των ουσιών είναι το πιο δύσκολο. σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Μην σοβαρότητα. Πρόεδρε, από ό,τι βλέπω κάνετε νόημα, όπω είπα, πολλά. Εάν θέλουν οι ε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, να του συζητήσουμε το θέμα, πολύ ευχαριστώ. Εάν δεν τους καλύπτουν οι απαντήσει μου. Ευχαριστούμε για την προθυμία σας κύριε Μέρφη. Σας ευχαριστούμε βαθέων για αυτές τις απαντήσεις. Γιατί πραγματικά έχουμε απελπιστεί. Έχουμε απελπιστεί σε μια Ευρώπη που τόσο πολλά ερωτήματα θέτουν ε, πολίτες για την αποτελεσματικότητά μας. Εδώ φαίνεται αισθανόμαστε σαν να προσπαθούμε να πρόξουμε έναν ογκόληθο για να πετύχουμε τέτοια πρόοδο. Θέλουμε λοιπόν ε, να δείξουμε στους Ευρωπαίους ότι η πρόοδος μπορεί να επιτελεστεί, ότι μπορούμε να ωφελήσουμε όμως και εκείνους και όχι μόνο την, ε, τον κλάδο. Ε, θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι όταν υπάρχουν σοβαρέ ανησυχίε μπορούμε να λάβουμε μέτρα. Ενώ συνήθω κάνουμε το αντίθετο τέλο πάντων. Λοιπόν, η αντίδρασή μου ως βουλευτού και κάποιων συναδέλφων φαντάζομαι και βλέποντα τι εκφράσει σα ε, εδώ στην αίθουσα είναι νομίζω ανάλογε. Σα ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ που ήρθατε. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, σημείο 22. παρουσίαση για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ για να μας παρουσιάσει την σχετική έκθεση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή το σημείο αυτό σίγουρα σας ενδιαφέρει πολύ, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κοινωνική και οικονομική έκθεση προέκυψε από αίτημα του Περιβαλλοντικού Συμβουλίου το Δεκεμβρίου 2008 για να διευνηθεί ο κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος της καλλιέργειας γαματαφόμικρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικές πληροφορίες ε, ήταν ε, ελλειπείς ή τελείως ανύπαρκτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν συγκέντρωσε τι απόψει των 100 μελών και των ενδιαφερομένων από τον Ιούλιο του 2009 και από τη μια καταστήσαμε σαφέ ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να υποβάλουν έκθεση ανα πάσα στιγμή εφόσον θεωρούν ότι υπάρχει κάτι εύστοχο που μπορούν να αναφέρουν. Και κατά τα άλλα, προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε, ώστε να επικεντρωθούν στα σημαντικότερα ζητήματα με ένα ενδεικτικό μάλιστα ερωτηματολόγιο που προμηθεύτηκε στα κράτη-μέλη από την Επιτροπή. Είχαν πάντως απόλυτη ελευθερία να μας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία ήθελαν. Αλλά έστω ενδεικτικά τους ζητήσαμε να μας πούν τα πιο σημαντικά, να μας εντοπίσουν τα πιο σημαντικά σημεία να πω ότι παρόλο που περιμέναμε ότι θα είχαμε πλήρεις και λεπτομερέστατες αντιδράσεις από τα κάτι μέλη, τελικά μόνο 25 απήντησαν. Δύο δεν απήντησαν καθόλου. Η Ιταλία και η Βουλγαρία συγκεκριμένα. Και επίσης είχαμε απαντήσεις από την Ορβηγία και άλλους ενδιαφερομένους. Άρα άφθονο υλικό για να το επεξεργαστούμε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι συμβολές των επιμέρους κρατών μελών απέκλειναν μεταξύ τους και ως προς την προσέγγιση και την ποιότητα και την τοποθέτηση. Κάποιοι είχαν μια μονοσέλιδη δήλωση, ενώ άλλοι ξεπέρασαν τις 200 σελίδες διεξοδικότατων μελετών και ενδελεχέστατων παρατηρήσεων. Κάποια κάτι μέλη για να απαντήσουν ετοίμασαν μια εθνική επισκόπηση, ενώ άλλοι προθέσεως απλώς ανέφεραν την ποικιλία απόψεων που υπάρχουν και μας τα σέρβιραν χωρίς επεξεργασία. Είχαμε λοιπόν ε, υλικό αρκετά αντιφατικό. Κάποιες πολύ ε, ε, ορθολογικές μάλλον και επεξεργασμένες απόψεις και κάποιες άλλες που ήταν σε ένα του τι συμβαίνει στον έξω κόσμο. Είναι σαφές και φυσικό να παρατηρήσουμε πόλωση των απόψεων στις συνεισφορές των κρατών μελών. Πραγματικά, αυτό στηρίχθηκε και από συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα Ευρωπαϊκής Εμβέλειας. Ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ε, η στήριξη με αποδεικτικά στοιχεία ήταν ε, Ελιπέστατη. Το φάσμα που καλύφθηκε ήταν πολύ ευρύ, παρόλα αυτά συνήθως υπήρχε αναφορά στο επίπεδο των ε, εκμεταλλεύσεων. Κάποια κράτη-μέλη που είχαν εμπειρίες τέλο πάντων από την καλλιέργεια γάματα φόμικρων όπως η Τσεχία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, η Σλοβακία και η Σουηδία ανέφεραν τα δικά τους εθνικά στοιχεία όπως την αύξηση των ε, ποσοτήτων ε, στη συγκομιδή με τις συγκεκριμένες καλλιέργειες. Ενώ άλλα κράτη-μέλη προφανώς επειδή δεν είχαν δικές τους εμπειρίες δεν μας ανέφεραν και τέτοια δεδομένα. Αρκετά κράτη-μέλη όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, οι κάτω και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και η Νορβηγία ήδη είχαν πλαίσια ανάλυση του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, βάσει των όσων προείπα, λόγω τη περιορισμένη διαθεσιμότητα και ποιότητα των στοιχείων και επειδή ήταν πολύ ετερογενή μεταξύ του, θεώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα ήταν άστοχο να περάσει σε λεπτομερέστερη ανάλυση αυτού του ετερογενού υλικού και να καταλήξουμε σε τελεσίδικα συμπεράσματα. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε κάποια από τα σημεία που θεωρήσαμε σημαντικότερα από όλες αυτές τις παρατηρήσεις ως ενάβσματα για να ξεκινήσουμε και να, να προτείνουμε κάποιες δράσεις. Επιπλέον, η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση της των ε, διεθνών επιστημονικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί και σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές διαστάσεις και όλη την κοινωνική αλυσίδα ή τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθήσαμε να ετοιμάσουμε μια διεξοδική παρουσίαση όλου του υλικού που είχαμε στα χέρια μας τη στιγμή της δημοσίευσης. Αυτό που προτείνουμε βασικά μετά από αυτή την ε, συλλογή πληροφοριών είναι να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε συζητώντα με τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερομένους, μήπως υπάρξει μια μετατόπιση. Από την πόλωση στις απόψεις, να βάλουμε αντικειμενικότερους στόχους στους εαυτούς μας. Νομίζουμε το πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε ένα στο σύνολο δικτών και παραγόντων. Γι' αυτό έχει ήδη δημιουργηθεί ομάδα εργασία με τη συνεργασία των κατών μελών, τη οποία η πρώτη συνεδρίαση προβλέπεται φέτο τον Νοέμβριο. Καλωσορίζω σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση και του βουλευτέ να συμμετάσχουν εφόσον το θέλουν. Έπειτα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορούμε την καλύτερη αντίληψη που θα έχουμε για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας γαματαφόμικρων να τις χρησιμοποιήσουμε και στην ίδια την καλλιέργεια και τη διαχείρισή της. Βάση για την επόμενη συνάντηση στην όλη διαδικασία που οργάνωσε ο Επίτροπος Ντάλι ο ίδιος θα είναι όλα αυτά τα υλικά που έχουμε συγκεντρώσει για το θέμα των γαματαφόμικων. 18 Οκτωβρίου, όπω θα έχετε ακούσει, θα συζητήσουμε σε μια πρώτη συνάντηση τα θέματα αυτά, κοινωνικέ και οικονομικέ επιπτώσει από την καλλιέργεια των γάμματαφόμικων. Πρόεδρε, σα καλωσορίζουμε και εσά, αφού σα ευχαριστήσω. Ε, σας καλωσορίζουμε, αν θέλετε, και να προεδρεύσετε σε μια από αυτέ τι συναντήσεις. Ε, αυτά ήταν τα στοιχεία που είχα να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ να απαντήσω στα ερωτήματά σα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Απλώ και εγώ να πω ένα μια σκέψη πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Η έκθεση αυτή που τόσο ανυπόμονα περιμέναμε με άφησε λιγάκι ανικανοποίητη. Διότι περιμέναμε να δούμε και την κοινωνική χρησιμότητα όλου αυτού του εγχειρήματο. Όχι μόνο τα οικονομικά στοιχεία, θέλαμε τα αρνητικά και θετικά στοιχεία από κοινωνική άποψη. Αυτό δεν το βρήκα στην έκθεσή σα ο κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος περιορίζεται στην αύξηση των εισοδοτημάτων και του κέρδους των γεωργών. Και μάλιστα μιας μερίδας των γεωργών. Διότι οι βιολογικοί καλλιεργητές, οι συμβατικοί, οι παραδοσιακοί τέλο πάντων γεωργοί, δεν λαμβάνονται καν υπόψη. Έχουμε λοιπόν την αίσθηση ότι στην έκθεση αυτή καλύπτεται ένα μέρος των επιστημονικών μελετών. Το θέμα αυτό υποθέτω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε επανειλημμένος. Γιατί δεν λάβατε υπόψη την αντίσταση που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στην ε, Λατινική Αμερική. Γιατί δεν λάβατε υπόψη όλου του φορεί τη αλυσίδα παραγωγή. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αντιμετωπιστούν με παρόμοια προσοχή. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Αρσένη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τεράστια σημασία στο θέμα των οικονομικών και κοινωνικών ε, επιπτώσεων της καλλιέργειας ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η Επιτροπή δηλώνει ότι χώρες όπως η Ισπανία καταγράφουν θετικές συνέπειες στην παραγωγικότητα σε περίπτωση προβλημάτων στις καλλιεργίες. Και ναι, μπορεί να υπάρχουν και επιχειρήματα ως προς την αυξανόμενη παραγωγικότητα το προϊόν, δηλαδή που προέρχεται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, που καταγράφει και η ίδια βιομηχανία, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε επιπλέον από ολόκληρο τον κόσμο μας με τις επίσημες έρευνες μάλλον τείνουν προς την αντίθετη διαπίστωση. Γι' αυτό και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας FAO έχει διατυπώσει ακριβώς το αντίθετο επιχείρημα ότι πρέπει, εάν θέλουμε να έχουμε ασφάλεια στην προμήθεια τροφίμων, αντίθετα από αυτό που υποστηρίζει η βιομηχανία, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς λιγότερο εντατική και προς παραδοσιακή δηλαδή καλλιέργεια και γεωργία. Μια άλλη μελέτη λέει ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε ότι για να προστατεύσουμε μάλλον τις παραδοσιακές ε, καλλιέργειες από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και την επιτυχία επιμόλυνση, χρειαζόμαστε ε, μια επιβάνηση κάπου στο 14%. Τελευταία απόφαση δε του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ανάγκη αποζημίωσης των μελισσοκόμων ε, που ε, πρέπει να καταβληθεί για την ε, επιμόλυνση των καλλιεργειών των φυτών από γενετικά τροπημένους οργανισμούς αποδεικνύει πόσο μεγάλο κόστος θα έχουμε για αποκατάσταση εφόσον δεν προστατεύουμε τις ε, παραδοσιακές μας ε, καλλιέργειες. Δηλαδή κινδυνεύει η ίδια, ο ίδιος ο πυρήνας της γεωργίας αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει ένα δρόμο ο οποίος θα μας οδηγήσει σε τεράστιο κόστος. Κόστος το οποίο θα πρέπει να καταγραφεί στο λογαριασμό των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η Επιτροπή μπορεί να απαντήσει, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, Σαντρίν Μπελιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει και εγώ να συμφωνήσω με την απογοήτευση που ξέφρασαν οι συνάδελφοι και να επισημάνω τα εξή. Δύο παρατηρήσει και δύο ερωτήσει στην Επιτροπή, όπου καταγράφεται το πότε και το τι και πότε και πώς. Για το πότε. Η πρώτη μελέτη αυτή για τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες της καλλιέργειας των γενετικά τροπημένων οργανισμών. Όμως έχουμε μια πρώτη αυτή από το ένα, θα έπρεπε, ε, μια πρώτη νομοθεσία. Το 2003 θα έπρεπε να έχουμε την πρώτη αξιολόγηση. Και έχουμε φτάσει το 2011 που μας ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα θεσπιστούν ομάδες εργασίας, ότι θα μελετηθεί η υπόθεση. 2011-2012 κανονικά θα έπρεπε να είμαστε στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης. Εδώ βλέπουμε μόλις την πρώτη. Και τώρα φτάνω στο τι και πώς. Προφανώς δεν είναι ε, η έκθεση αυτή στο ύψος των περιστάσεων. Δεν δίνει απαντήσεις. Έχουμε όλες αυτές τις σελίδες οι οποίες δεν έχουν καμιά ουσία, είναι κενές περιεχομένου, δεν δίνουν καμία απάντηση, δεν μας καθεσυχάζουν ως προς τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες των γενετικά τροπημένων οργανισμών και τη στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Δεν υπάρχει παρά μόνο μια, ένα συμπίλημα πληροφοριών χωρίς αντικειμενικότητα, χωρίς κατευθυντήριες γραμμές, ε, χωρίς μέθοδο. Ένα κείμενο δηλαδή το οποίο δεν μας προσφέρει τίποτα και δεν μας λέει τίποτα. Ερωτώ λοιπόν και πάλι στο πότε. Πότε θα έχουμε εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση που να αξίζει και τον τίτλο της έκθεσης με αξιολόγηση των συνεπειών της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και όπως είπαμε, όχι μόνο με την οπτική γωνία του καλλιεργητή της γενετικά τροποποιημένης ε, του γενετικά, γενετικά τροπημένου οργανισμού, αλλά τις συνέπειες στα τρόφιμα, τις συνέπειες για τον καλλιεργητή της παραδοσιακής καλλιέργειας, για τον καλλιεργητή της βιολογικής Καλλιέργεια κοινωνικο κοινωνικο-οικονομικά, τι συνέπειες σημαίνουν, ε, ε, επέχουν αυτές οι γενετικά τροπημένοι οργανισμοί προ τη δημιουργία της τι την επιβίωση της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος κερδίζει από του γενετικά τροπημένου οργανισμού, η γεωργία κερδίζει, η ε, γεωργική χημεία, η βιομηχανία των τροφίμων, ποιο κερδίζει από όλα αυτά και επίση καλό θα ήταν να μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να ξέρουμε τι είδου γεωργία διαλέγουμε, τι είδου προϊόντα θέλουμε να προσφέρουμε στον Ευρωπαίο ε, πολίτη. Όλα αυτά τα στοιχεία τα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να λάβουμε σε αποφάσει. Αυτά ήταν τα πώ λίγο πολύ, ελπίζοντα ότι ε, θα έχουμε σχετικά σύντομα αυτή τη μελέτη με απαντήσεις ε, σε όλα αυτά τα ερωτήματα και επίση πρέπει να πω ότι αισθάνθηκα κατάπληξη από ένα από τα στοιχεία της εκθέσεως που λέει ότι θεωρείται εφικτή η συνύπαρξη μη, γενετικά τροποποιημένων και γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Δηλαδή, μας λέτε ότι είναι δυνατόν να παραμείνουν καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένες μαζί με μη γενετικά τροποποιημένες. Εάν είναι έτσι, τι έχετε να πείτε για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον Ευρωπαίο Μελισουργό που καταγράφει ξεκάθαρα ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συνύπαρξη γενετικά τροπημένων οργανισμών και κυρίως το 810 με την ε, μελισσουργία, μελισσοκομεία. Ο κύριος Στάσα, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Με προσοχή διάβασα αυτή την έκθεση και μπορώ φυσικά να προσθέσω και τη φωνή μου στα σχόλια των προλαλισσάντων. Ειλικρινά δηλαδή. Αυτά τα οποία διαβάζει κανείς σε αυτές τις 11 σελίδες είναι πολύ απογοητευτικά. Είναι Απογοητεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ομολογεί κατά το μάλλον ή ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι φαίνεται ότι αντέγραψε μόνο στοιχεία τα οποία απέστειλαν τα κράτη-μέλη. Θα έπρεπε να γίνει μια περαιτέρω ανάλυση όμως σε σχέση με τις απαντήσεις και τα στοιχεία αυτά. Κάτι να υπάρξει σε σχέση με την συλλογή αυτών των στοιχείων που δεν είναι ιδιαίτερα πιστική αυτή η συλλογή, η σταχειολόγηση στοιχείων. Ένας κατάλογος απόψεων ή στοιχείων ε, μπροστά σε μια ε, κατάσταση που έχει πολλωθεί και όσον αφορά και την βιβλιογραφία για τις ε, επιπτώσεις και για τα γενετικά τροποποιημένα. Ποιο είναι το όφελος όλων αυτών και ποια μέθοδος βρίσκεται πίσω από τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ποιος είναι ο στόχος και η δομή μεθοδολογικά. Θα έπρεπε καταρχήν να προσδιοριστεί ως ορισμός ποιε είναι οι επιπτώσεις όλων αυτών. Και πολύ σωστά αναφέρθηκε από σχόλιο που ακούσαμε προηγούμενα, είναι υπερβολικά μονοβαρής, μονόπλευρη η προσέγγιση και πουθενά δεν βρίσκεται και σε αυτή την έκθεση το στοιχείο ότι για παράδειγμα σε σχέση με τα γενετικά τροποποιημένα στην Ισπανία που αναφέρεται ότι σε τρεις επαρχίες οι γεωργοί εκεί λέει έχουν μεγαλύτερη σοδιά 8, τόσο Εξαιρετικό, τέλεια. Όμως θα έπρεπε να δούμε ότι αυτή η μεγαλύτερη σοδιά αναφερόταν μόνο σε αυτές τις τρεις ε, επαρχίες. Τέλεια, εξαιρετικά. Τι σημαίνουν όλα αυτά και τι συνεισφέρουν όλα αυτά σε μια τέτοια έκθεση. Ποιο είναι το όφελος. Καθόλου δεν είναι σαφές ποιες κοινωνικές οικονομικές επιπτώσεις υπάρχουν από τα γενετικά τροποποιημένα Λοιπόν, γιατί πάντα και μόνο αναφέρεται το θέμα των ίδιων των γεωργών ατομικά. Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν όμως σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων. Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν στους συμβατικούς γεωργούς και στους βιογεωργούς βιολογικής, βιολογικών καλλιεργειών. Και αυτά τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο αυτής της εικόνας ε, ως ε, συνόλου. Και να μην αναφερόμαστε μόνο ατομικά σε κάποιους γεωργούς που καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένα Τώρα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μικρότερη ύπαρξη τέτοιων καλλιεργιών στην Ευρώπη, ενώ υπάρχουν πολύ περισσότερες στις ΗΠΑ και εκεί πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία. Ακόμα και μικρής έκτασης ε, γενετικά τροποποιημένων, ακόμα και στους μικρότερους γεωργούς. Να δούμε τις επιπτώσεις. Και διαβάζω και κάποιες επισημάνσεις σε αυτές τις 11 σελίδες, ισχνές και παρατηρώ ότι πρόκειται για σταχειολόγηση. ένα ανθολόγιο ουσιαστικά που έχει επιλεγεί από την βιβλιογραφία και τα επιστημονικά στοιχεία. Πολύ μονομερός, πολύ μονοβαρός. Αναφέρεται η περίπτωση του Graham Brooks. Είναι εκείνος ο οποίος είναι επικεφαλής του γραφείου ε, ε, Economics και έχει παραγγελίες σε σχέση με την ε, βιογεωργία. Αν αυτό το προσκομίσει κανείς ως στοιχείο Πού βρίσκεται η αμεροληψία και πού βρίσκεται η αντικειμενικότητα της επιστημονικής προσέγγισης και έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να προσθέσω το σχόλιο μου στο σχόλιο της κυρίας Μπελιέ. Τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα, υπερβολική καθυστέρηση υπάρχει σε σχέση με τα όσα κάνουμε. Πώς θα καταλήξουμε στα στοιχεία και τα συμπεράσματα τα οποία απουσιάζουν μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. And uh, Σε ευχαριστούμε. Κυρία Λεωτάρ τώρα παρακαλώ. Yeah, Σε ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου στα σχόλια των προηγούμενων αγοριτών. Στο Συμβούλιο για τα θέματα περιβάλλοντος του 2008 ζητήθηκε να υπάρξει μια αξιολόγηση πριν από τρία χρόνια, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, τώρα, σήμερα, έχουμε μια τελείως αναδιαρθρωμένη συλλογή στοιχείων από τα κράτη-μέλη που μας παρουσιάζεται και αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εξειδικευμένη ομάδα γεωργών και τα οικονομικά τους ε, ε, έσοδα. Αυτό που λείπει όμως είναι η περίπτωση της ε, βιοπικιλότητας, η επίπτωση για την απασχόληση. Τι γίνεται με τα αναπτυσσόμενα κράτη και κατά πόσον η ευρωπαϊκή ρύθμιση αυτή έχει επιπτώσεις για παράδειγμα όσον αφορά την καλλιέργεια σόγιας στη Νότια Αμερική και ποιες επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στον τομέα των τροφίμων. Τι επιθυμούν οι καταναλωτές, τι επιθυμούν σε σχέση με τις βιοκαλλιέργειες. Όλα αυτά δεν ελήφθησαν υπόψη και απουσιάζουν. Διερωτώ με λοιπόν, τι θα κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θεματικό πλέγμα. Πώς θα το προσεγγίσουμε, ποιοι ανεξάρτητοι επιστήμονες θα αξιολογήσουν αυτά τα κοινωνικά οικονομικά στοιχεία, ποιο θα είναι το κέντρο βάρους σε αυτή την αξιολόγηση, την εκτίμηση που πρόκειται να γίνει και πώς όλα αυτά, αυτή η εκτίμηση, η αξιολόγηση θα ερμηνευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, οι κοινωνικο-οικονομικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις είναι κάτι για το οποίο αναμένουμε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, απογοητευτικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και συνεχίζουμε να έχουμε νέες ε, προδιαγραφές και διατάξεις για την αντιμετώπιση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων ε, χωρί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι κοινωνικονομικές πτυχές και Χωρί χωρίς ε, καν να υπάρχουν σημεία σημείο αναφοράς. Και υπάρχουν εδώ και ρυθμίσεις σχετικά με τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Αυτά όμως οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις δεν, ε, δεν εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο και δεν αφομοιώνονται. Τι θα κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά στο μέλλον. Αυτά είναι πρόσθετα ερωτήματα στα οποία, ε, σε εκείνα τα οποία διατύπωσαν οι συνάδελφοι πιο πριν. Ευχαριστούμε. Ούτε εγώ βρήκα πολύ ικανοποιητική την έκθεση αυτή. Έχω όμως να θέσω κάποια ερωτήματα στους ε, εκπροσώπους της Επιτροπής. Εφόσον μιλάμε για επιπτώσεις κοινωνικές και οικονομικές, γιατί δεν έγινε αναφορά στα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για την Αμερικανική βιομηχανία ρυζιού, παραγωγής ρυζιού. κυρίως για την αγορά γενετικώς τροποποιημένου ρύζιου από την Μπάγκερ που έφτασε ως την Ευρώπη. Επίσης υπάρχει μελέτη από την καθηγήτρια Μπινιμέλης που αναφέρει ότι στην Ισπανία μειώθηκε κατά 2 τρίτο αριθμός βιολογικών γεωργών και καλλιεργειών λόγω της μόλυνσης από τους γενετικώς τροποποιημένε καλλιέργειες. Γιατί επίση δεν αναφέρεστε στο γεγονό ότι οι πολυεθνικές πολλούν σπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως εταιρείε που έχουν ε, καταγγελθεί από μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως η Μονσάντο. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά. Επίσης γιατί δεν λέτε ότι επιβάλλονται στους εισαγωγείς, τους εξαγωγείς, τους παραγωγούς και τους καλλιεργητές οι καλλιέργειες αυτές και τους αφήνονται πολύ λίγες δυνατότητες για να κρατήσουν ελεύθερες από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς τις καλλιεργίες τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σώρευση στοιχείων και δεδομένων και αυτό που κυρίως με εκπλήσει είναι ότι η έκθεση παρουσιάζει ως επιτυχίες την καλλιεργία την καλλιέργεια του αραβοσίτου 810 Μονσάντο στην Ευρώπη, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τσεχία. Αλλά τα κέρδη δεν είναι τόσο σοβαρά και καθόλου δεν αναφέρεται η μελέτη της Τσεχίας μεταξύ των καλλιεργητών Μονσάντο 810. Ούτε υπάρχει μνήμα καμιά επιστημονική μελέτη που να δημοσιεύτηκε σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό, έτσι. Αναφέρονται τρία άρθρα τα οποία έχουν ε, συνταχθεί από τον ε, κύριο Μπρούκερς, ε, που είναι ένας από τους γνωστότερους επερασπιστές της γενετικώς τροποποιημένης βιομηχανίας και αυτό σε φόρουμ το οποίο χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και τη σχετική βιομηχανία. Επίσης, επί τριετία, η συγκομιδή από τις καλλιέργειες αυτές ήταν χαμηλότερη από μάλλον ήταν ανώτερες από τις παραδοσιακές και βιολογικές μορφές καλλιέργειες, αλλά λέγεται σε αστερίσκο στο κάτω μέρος της σελίδας ότι ήταν τυχαίο το γεγονός αυτό και δεν είναι αξιοποιήσιμο στοιχείο. Επίσης η έκθεση αναφέρεται σε περάτωση σχεδίου, του σχεδίου Ιδίω όταν οι τα γενετικώ τροποποιημένα προϊόντα θα βρίσκονται στα ράφια των ευρωπαϊκών καταστημάτων, θα τα αγοράζουν οι καταναλωτέ. Αναφέρεται όμω ότι στα αγγλικά σούπερ μάρκετ δεύτερη κατηγορία κάποια από τα έλαια που. λέγεται στην ετικέτα, δεν λέγεται στην ετικέτα τους ότι περιέχουν ε, γενετικώς τροποποιημένα συστατικά, αγοράζονται από τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Και για την εμπορία των προϊόντων αυτών σε μια περιοχή κοντά στη δική μου, στο Φρίουλι Βενέτσια Τζούλια. Δεν φαίνεται να έγινε να ήταν μεγάλη επιτυχία του γενετικώς τροποποιημένου του Τέλος πάντων, αναφέρω την Ιταλία γιατί εμείς δεν απαντήσαμε στο ερωτηματολόγιο όπως ε, μόνο η Βουλγαρία έκανε. Εντάξει, εσωτερικές υποθέσει αυτές θα μου πείτε, όλοι τις καταλαβαίνετε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρέιμερς. Um, σας, ευχαριστώ. Βλέπει κανείς ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημα. Ένα δίλημα κατά τούτο, μια και πρέπει να διαπιστωθεί ότι συντάσσοντας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτες που εξαρτώνται από τα στοιχεία των κρατών μελών με πολύ διαφορετικό τρόπο, τρόπο και βάθος και τελείως διαφορετική αξιολόγηση χρησιμοποιούνται αυτά. Το επόμενο στοιχείο. Θέλουμε ένα σημείο, ένα θέμα αντικειμενικά, με αντικειμενικό τρόπο να τα συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε κάθε μελέτη που συντάσσεται ως αντικειμενική όταν προέρχεται από τους οικονομικούς κύκλους. Θα πρέπει όμως από τις ε, περιβαλλοντικές ομάδες ε, οι αντίστοιχες μελέτες πώς να βαθμολογηθούν, υποκειμενικές, τουλάχιστον θα πρέπει με ένα δίκαιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τις ε, διάφορες μελέτες και αξιολογήσεις. Θα με ενδιαφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μελέτη για τις κοινωνικές οικονομικές επιπτώσεις αυτών των καλλιεργειών, κατά πόσον να δούμε ποιες επιπτώσεις υπάρχουν στην Ευρώπη αν χρησιμοποιείται αυτή η καλλιέργεια ή όχι και να δούμε η Ευρώπη όντας ε, για παράδειγμα το τελευταίο οχυρό παγκόσμια όπου ε, δεν αναγνωρίζονται αυτές οι μέθοδοι και να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν εκτός Ευρώπης να ρυθμίζεται η συνύπαρξη των ε, καλλιεργιών αυτών χωρίς να αποβαίνουν εις βάρος των βιοκαλλιεργιών και να καταλήξουμε σε μια αντικειμενική βάση. Δεν είναι το θέμα το αν είναι κανείς υπέρ ή κατά τέτοιων καλλιεργειών, αλλά ως πολιτικό θεσμικό όργανο, ως Ευρωκοινοβούλιο, θα έπρεπε με αντικειμενικό τρόπο, σε αντικειμενικά στοιχεία να βασιζόμαστε σε αυτή τη συζήτηση και λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένοι να τα συζητούμε. Αυτό να μένουν και οι πολίτες, αντικειμενικά να τα συζητούμε και όχι με ε, φορτισμένοι συγκινησιακά να τοποθετούμαστε. Και εδώ πραγματικά πρέπει πρέπει να πούμε ότι πολύ έντονα υπάρχουν συναισθηματικού χαρακτήρα επιχειρήματα και πολύ λιγότερο με βάση αντικειμενικά στοιχεία γίνεται αυτή η αντιπαράθεση. Ήρθε επιτέλους η χρονική στιγμή να καταλήξουμε σε αποφάσεις που θα λάβουμε και όχι με βάση τέτοιων συζητήσεων που ε, έχουν επιβαρυνθεί ε, συναισθηματικά διότι η Ευρώπη δεν είναι μόνη της στην παγκόσμια σκηνή. Υπάρχουν και άλλες χώρες και άλλες ήπειροι. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Τώρα, άσχετα από το γεγονός ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο και χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο εύρος προσέγγισης για τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχα κάπως την εντύπωση που αποκόμισα ότι κάπως σας εκπλήσει ότι δεν υπήρχε κάποιο σαφές αναμφίσιμο αποτέλεσμα σε σχέση με αυτή τη μελέτη. Αν δει κανεί τη, γραμμή αφετηρία ουσιαστικά εθελοντικά, εθελούσια μπορούσαν τα κράτη-μέλη να αποστέλουν πάσης φύσεως στοιχεία προς εμάς. Και στο τέλο δεν πρέπει να εκπλήσεται κανείς ότι όλα αυτά δεν βρίσκονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Θα ήθελα να, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω το εξή. Υπάρχει η φόρτιση η συναισθηματική, ότι δηλαδή εσκεμμένα αφέθηκαν τα τρία χρόνια να περάσουν για να μην καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα το οποίο θα δυσαρεστούσε ίσως σε κάποιους βιομηχανικούς κύκλους. Εγώ θα χαιρόμουν αντίθετα αν δεν αφήνατε το χρόνο να περνάει, αλλά κάποια από τα θέματα που τέθηκαν από τους με πιο ικανοποιητικό τρόπο θα προσπαθούσατε να καλύψετε και να απαντήσετε σε αυτά. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Ο κύριος πρώτη τελευταίος αγορητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπούμε που στο κείμενο δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές της ε, έρευνες της γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να δώσει περισσότερη ουσία στην συζήτησή μας. Ε, στο θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, νομίζω πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι, πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορούμε να εμβαθύνουμε. Και να είμαστε πάντα ε, προσεκτικοί, να ακολουθούμε την αρχή της προφύλαξης. Γιατί μια τροφή γενετικά τροποποιημένη δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής για την υγεία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα δούμε εις βάθος και να έχουμε μία βάση αναφοράς για το μέλλον. Έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε την καταλληλότερη λύση. Σήμερα πρέπει να οργανωθούμε, ακόμα και με τη βοήθεια της ΤΟΑ, και να έχουμε μια συζήτηση λεπτομερέστατη για αυτό το θέμα. Εγώ προσωπικά έχω την τάση να θεωρώ ότι δεν είναι αναγκαστικά επιζήμια για τον οργανισμό οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί και αυτοί. Υπάρχουν όμως ενδεχομένως επιπτώσεις. Το έχω θίξει και στο παρελθόν στη συζητήση της Επιτροπής, μου, της μας. Επιπτώσεις που με κάνουν να διερωτώ γιατί τέτοια πίεση για τη χρήση σπόρων και σπορών γενετικώς τροποποιημένων. Μπορεί να είναι μόνο η βελτίωση στη συγκομιδή, στη σοδιά ο στόχος. Ακόμη και όταν αυτό είναι επιτυχές ως προσπάθεια, είναι επικίνδυνο ταυτόχρονα, διότι θα εξαρτήσουμε την ε, διατροφή του πλανήτη μόνο σε λίγες φυτικές ποικιλίε και καλλιέργειες που θα μπορούσαν κάποια στιγμή να κινδυνέψουν ε, αν υπάρξει λόγω χάρη κάποια επιδημία ζυζανίων ή άλλου είδους. Η περιορισμένη λοιπόν επιλογή σπόρων, εφόσον μπορεί να υπάρξει μία επίθεση κατά της συγκεκριμένη ποικιλία, θα είναι καταστροφική για τις δυνατότητες θρέψης και ολόκληρης ανθρωπότητας. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία καλό θα ήταν λοιπόν να τα σκεφτούμε. Μαζί και με το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει να κάνει με τις καλλιέργειες αυτές. Όλα αυτά μπορεί να μας βλάψουν εάν δεν υπάρχει έστω και ελεύθερη χρήση αυτών των ποικιλιών. Ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό το τελευταίο στοιχείο που αναφέρατε. Πράγματι, όταν υπάρχει σπορά σπόρος που προστατεύεται από δίπλωμα βιστεχνία, τότε αυτό επηρεάζει και την τιμή. Έχω και εγώ δύο σύντομα σχόλια. Στη σελίδα 8 λέγεται ότι ο καταναλωτής, μάλλον οι καταναλωτές, όταν απαντούν στα ερωτηματολόγια αν θέλουν να αγοράσουν γάματα φόμικρον ή όχι, λένε ότι δεν έχουν πληροφορίες αν τελικά τα αγοράζουν ή όχι. Δύσκολα. Ε, περίεργη δεν είναι η διατύπωση εδώ. Γιατί δεν λέτε ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι κατά οι καταναλωτές. Εκεί θα είχαμε πολύ καλύτερες, πολύ πιο αξιόπιστες πληροφορίες. Και κάποιε φορέ όταν βιάζεται κανεί να ψωνίσει στο κατάστημα, δεν κοιτάει και με τόσο μεγάλη προσοχή την ετικέτα. Επίση, λέτε ότι το καθαρό κέρδος, περιθώριο κέρδο για του ε, καταναλωτέ τη Αργεντινή είναι σοβαρό Υπάρχει τέτοιο περιθώριο, διότι εγώ άκουσα το ακριβώ αντίθετο, ότι είναι τόσο ανθεκτικό το σιτάρι, ο σίτος που καλλιεργούν εκεί πέρα, που χρειάζεται να αγοράζουν όλο και περισσότερα ζανιοκτώνα ετησίως. Και τελικά είναι πολύ ε, αναποτελεσματική η καλλιέργεια αυτή. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά ερωτήματα για να απαντήσετε σε όλα αυτά, αλλά μην το ξεχνάμε, το αρχικό ερώτημα ήταν η απόφαση του ΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μάλλον. Το θέμα της... του μελιού και της μελισσοκομείας. Μπορείτε να απαντήσετε και γι' αυτό. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε όλα. Και για το μέλι και για την απόφαση του δικαστηρίου. Να αντιδράσω πολύ σύντομα σε τόσο πολλά σχόλια που ακούσαμε και τόσες πολλές ερωτήσεις. Δεν μπορώ ένα προς ένα να τα απαντήσω. Είμαι όμως ανοιχτός. Όποτε θέλετε να συναντηθούμε. Να τα πούμε με λεπτομέρειες, εφόσον τόσο πολύ σας ενδιαφέρει το θέμα. Σας καλώ και στη διάσκεψη στις 18 Οκτωβρίου, όπου ακριβώς με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε, με όλους τους τομείς που αναφέρατε εδώ. Γι' αυτό άλλωστε την οργανώνουμε τη διάσκεψη αυτή ώστε όλες οι πλευρές να ακουστούν, όλες οι απόψεις συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, του μηχανικού κλάδου και το καθεξής. Ελπίζω ότι εκεί θα έχετε περισσότερες και βαθύτερες πληροφορίες. Είπατε επανειλημμένος, τέλος πάντων συχνά, αυτό που δέσποζε εδώ στη συζήτηση είναι ότι απογοητεύεστε, έχετε απογοητευτεί από την έκθεση. Σε αυτό πρέπει να απαντήσω. Γιατί όταν εξετάζαμε το θέμα στην Επιτροπή, είχαμε ήδη αξιολογήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες με Έναν στόχο όμως τον οποίο πρέπει να τον στηρίξουμε λογικός και επιστημονικός. Πριν ξεκινήσουμε τη μελέτη, πρέπει να ξέρετε ότι πολλά κρατημέλη τι μας έλεγαν. Έχουμε πολλές πληροφορίες, θα σας δείξουμε εμείς τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό που αναφέρεται εκεί, το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό, έχουμε να σας τα πούμε, αλλά όταν τα ζητήσαμε επισταμένως και συγκεκριμένα, τι πήραμε. Κοιτάξτε τις εκθέσεις των κρατών μελών. Το υλικό επισήμως τα κάτι μέλη το στέλνουν στην Επιτροπή. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ακούστε να δείτε Ισπανία λέτε ότι να είναι. Είναι επίσημες πληροφορίες της Ισπανίας αυτές. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τα διασταυρώσαμε με τα δημοσιευμένα στοιχεία, αλλά Είδαμε τα άρθρα και τα δημοσιεύματα τα οποία ήδη υπήρχαν σε άλλες πηγές, τα συγκρίναμε, τα αντιπαραβάλαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, είδαμε ότι οι ΜΕΝ και οι ΔΕ είναι, έχουν τεκμηριωμένα στοιχεία, δεν μπορούσαμε να πάμε παραπέρα προς την αξιοπιστία. Αυτό λοιπόν που μπορώ να πω προσωπικά οπωσδήποτε είναι ότι και εγώ απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα τις πληροφορίες που μου στείλανε δεν ήταν στο επίπεδο των προσδοκιών μου. Άλλα περίμενα από τα κράτη-μέλη, άλλα μας λέγανε πριν. Εμείς φανταστήκαμε ότι θα είχαμε μια χιονοστιβάδα πληροφοριών που θα μας πλακώσει. Και τελικά ήταν πολύ λίγα αυτά που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί. Στείλτε μας και άλλα στοιχεία. Ευχαριστώ. Αλλά πρέπει και να τα μπορούμε να τα κυρώσουμε και επιστημονικώς να είναι έγκυρα και να τα έχουμε διασταυρώσει. Είμαι πάντως ανοιχτό σε κάθε συζήτηση. Τώρα, αφού συγκεντρώσαμε το υλικό, αφού συντάξαμε την έκθεση, προέκυψαν και κάποιες νέες πληροφορίες. Ε, βεβαίως και τα χρησιμοποιήσαμε και αυτά. Καθώς εξελισσόταν η διαδικασία, φροντίσαμε να τα ενσωματώσουμε. Θα γίνει αυτό και με τη διαδικασία που ξεκινάει στις 18. Το κάναμε και τα αποστήλαμε και στο κοινό κέντρο έρευνας και θα συνεχίσουμε να τα συμπεριλαμβάνουμε στις εκθέσεις. Βασιζόμαστε όμως στις πληροφορίες που μας διέθεσαν άλλοι. Uh, which, which I won't probably... one... Υπάρχουν ε, πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά σας μένει ένα λεπτό. Καλά λοιπόν, θα σας μιλήσω για το μέλι. Τα υπόλοιπα άλλη φορά. Η απόφαση του δικαστηρίου για το μέλη λοιπόν. Η κατάσταση πραγματικά είναι σοβαρή. Ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ να ετοιμάσει γνωμάτευση για την ασφάλεια της ε, γύρης πώς μπορεί να επηρεαστούν τα προϊόντα μελιού. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έγκριση για συγκεκριμένες ουσίες ε, για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερη γραμμή για το μέλι. Για τη γύρη μάλλον. Αυτό θα πρέπει να έχει διατεθεί λογικά ως τον Οκτώβριο. Ζητήσαμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη και τις εταιρείε να κάνουν ό,τι μπορούν για να πληρωθεί το υπάρχον ρυθμιστικό κενό σε σχέση με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει εδώ να καλύπτεται κάθε φάσμα οποιοδήποτε διατροφικής χρήσης της γύρης υπό την έννοια του ισχύοντο ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα, αλλά από κοινό με τα κράτη-μέλη εξετάσαμε και τι υπόλοιπε πτυχέ. Το ζήτημα είναι πώ αξιολογεί κανεί την ετικέτα. Τι πρέπει να γράφει. Γύρι, στοιχεία ε, γενετικώ τροποποιημένα στη γύρι και μετά στο μέλι ή κατευθείαν στο μέλι. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε σε σχέση με το τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Από τη δική μας την πλευρά μπορώ να πω απλώς ότι ο Επίτροπος Νταλή τα θέματα αυτά θα τα αναπτύξει πλήρως στην Επιτροπή Γεωργίας. Καλώς, αλλά δεν θέλει ο μελισσουργός του ή να έχει τέτοιο, τέτοια γύρι στο μέλη του. Και θα πρέπει την επιβάρυνση αυτή, τη ζημιά που υφίσταται δηλαδή ο μελισσουργός, να την πληρώσει αυτός που έβαλε τη σχετική γύρι. Δεν μπορεί να μας επιβάλλει κανείς τέτοιου είδους προϊόντα. Πρέπει να το συστήσουμε αυτό. Λοιπόν, το πράγμα το έχει λήξει η συνεδρίαση και δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Γκεμπράντι για την επίσκεψή του. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο oh. ακόμα. Οι διερμηνείς τι λένε. I'm listening to Swedish. If I listen to English, could they inform me? Is it okay? Three more minutes? Okay, thank you. Uh, please, Jan. Um, Ευχαριστώ, Καρλ. Θα τα πω αγγλικά για να είναι τα πράγματα πιο απλά. Όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε το πρωί είχαν να κάνουν με επιστημονικά δεδομένα, πληροφορίες και το καθεξής. Αυτό είναι και η πεμπτουσία της, του δικού μας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Περιβάλλον. Πολύ σύντομα λοιπόν να πω ότι συζητήσαμε κατά την επίσκεψή μας πριν από λίγες εβδομάδες με την επίσημη αντιπροσωπεία όπου συμμετείχαν ο κύριος Σόνεκ, ο κύριος Ασένης και εγώ ίδιος. Υπήρχαν και μερικοί δανείς συνάδελφοι που ήρθαν μαζί μας. Η κυρία Ρόσπαχ. Τέλος πάντων μια σεβαστή αντιπροσωπεία. Στον κύριο Φούξ και τον κύριο Μπαζά ήθελα να του ευχαριστήσω για το έργο του από την πλευρά τη Γραμματεία. Ήταν τέλεια διοργανωμένη η επίσκεψη. Και πέραν του οργανισμού είχαμε και ένα επίσημο γεύμα στο Δανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όχι με τον ίδιο τον Υπουργό βέβαια, λόγω των εκλογών, αλλά με κάποιους από τους υπαλλήλους του Υπουργείου, συζητώντας τις προθέσεις της επερχόμενης Προεδρίας. Πολύ σύντομα να διατρέξω τα θέματα που θίξαμε. Με μεγάλη χαρά ε, ακούσαμε τον διευθυντή Τζάνετ Ματκλέιντ που ήταν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης την διευθύντρια μάλλον, ε, η οποία είναι μια από τις κινητήρε μου και μας είπε ότι ο οργανισμός προσπαθεί να χρησιμοποιεί κανονικούς ανθρώπους στο δικό τους φυσικό περιβάλλον για να συλλέγει τα δεδομένα του. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν ότι τις πληροφορίες του οργανισμού προφανώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όπως για τα επιθετικά είδη και ούτω καθεξής. Ε, ο οργανισμός πρώτος ο ίδιος μάλλον ο καλλιεργητής είναι ο πρώτος που θα εντοπίζει αν κάτι πάσχει από κάποια ασθένεια έχει μολυνθεί και είναι πολύτιμη συνεισφορά του οργανισμού όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει επίση στήριξη από ιδιώτε δωρητέ. Κάτι ακόμα που συζητήσαμε με τον οργανισμό είναι τα θέματα τη βιοπικιλότητας και κάποιοι οι του οργανισμού μας είπαν ότι υπάρχουν κενά στη βάση δεδομένων. Χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη γραμμή σύλλογης δεδομένων για την βιοπικιλότητα και αυτά αναφέρονται και στα δημοσιεύματα του οργανισμού. Λόγω έλλειψης χρόνου λοιπόν δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Συζητήσαμε τις κλιματικές αλλαγές και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού της ατμόσφαιρας. Για τις κλιματικές αλλαγές ξέρετε ότι είχαμε την έκθεση ΧΑΟΚ πρόσφατα με περισσότερα κονδύλια για τον οργανισμό καθώς και την ε, απόφαση για την κατανομή των ε, προσπαθειών. Θα πρέπει να εκτελεστεί από τον οργανισμό που θα έχει περισσότερη δουλειά λοιπόν και πολλές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό προβλέψαμε ήδη ένα επιπλέον κονδύλι. Ελπίζω να το εγκρίνει και ολομέλεια. Για την ε, ποιότητα της ατμόσφαιρας, νομίζω το πλέον ενδιαφέρον είναι ότι τα κάτι μέλη έχουν καθυστερήσει υπερβολικά ως προς την υλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Πάντως, σύμφωνα με τον οργανισμό, υπάρχουν ε, σοβαρότατοι λόγοι να έχουμε ακόμη αυστηρότερους κανόνες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, το ατμοσφαιρικό αέρα. Ένα σκληρός λοιπόν αγώνας προβλέπεται τα επόμενα χρόνια. Και άλλα Πάρα πολλά έχω. Ναι, αλλά οι Γερμανοί μου δώσαν τρία λεπτά. Τέσσερα άκουσα εγώ, είμαι στα τρισήμιση. Προχωράω στην ε, ε, αποτελεσματικότητα των πόρων. Δεν θα περάσω σε λεπτομέρειε, αλλά από τη δική του πλευρά έχουν ετοιμάσει προφίλ αναχώρα για το σημείο αυτό και μα είπαν ότι η αποτελεσματικότητα των πόρων γίνεται προτεραιότητα για τα περισσοτερα κατημέλη πλέον. Όμω ε, τα οικοσυστήματα και οι υπηρεσίε για τα οικοσυστήματα είναι κάτι που είναι τελείω ξεχασμένο. Κανεί δεν δίνει διάρα γι' αυτό. Τέλος, να καλέσω τους συναδέλφους να αξιοποιούν τον οργανισμό. Αν είναι κανείς εισηγητής, με πολύ μεγάλη ευκολία μπορεί να, επαφή, να έρθει σε επαφή μαζί τους. Πάρτε τηλέφωνο, ζητήστε τους να έρθουν εδώ ή να πάτε εσεί εκεί. Είναι πολύ απλό. Και μπορείτε έτσι να κάνετε την έκθεσή σας πολύ καλύτερης ποιότητας από ό,τι είναι συνήθω οι εκθέσει μα. Τελική παρατηρήση, Πρόεδρε. Μέχρι το τέλο τη χρονιά πρέπει να διορίσουμε νέο εκπρόσωπο από το δικό μα το Κοινοβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Είναι μια τριετή θητεία, η θητεία αυτή, και νομίζω ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου καλό θα ήταν να έχουμε σκεφτεί υποψηφίου. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να μας δώσουν ονόματα ανθρώπων που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν σωστά το Κοινοβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Συγκεκριμένε πληροφορίε μπορείτε να βρείτε και από του συναδέλφου του κ. Μπαζάν και Κρήτονα, 10 και χωρί διερμηνία. Έχουμε πάρα πολλέ πληροφορίες από τον οργανισμό για όλα τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα, το του ταφόμικρο, τους διαδράκτε, του τους ε, Λυπάμαι που έχει φύγει η Επιτροπή, θα το τους το ξαναπώ. Ας χρησιμοποιούν και εκείνοι τους πόρους του οργανισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Λυπούμε που καθυστερήσαμε τόσο. Τελική παρατήρηση